<laughs> Okay, friends, we'll start Καλημέρα φίλοι. Ας αρχίσουμε για να μπορέσουμε να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα ε, της ψηφοφορίας. Ε, σημείο πρώτο, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Νομίζω ότι μπορούμε να την εγκρίνουμε χωρίς τροποποίηση, έτσι δεν είναι. Yes, we can. Θυμίζω ότι το απόγευμα θα αρχίσουμε στις 3 και όχι στις 2.30 όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά. Ε, σημείο 2. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Διερμηνία έχουμε σε όλες τις γλώσσες με εξαίρεση τα σιουηδικά και τα κροατικά. Δεύτερη ενημέρωση. Συνεδρίασαν οι συντονιστές μας τελευταία φορά 12 Ιουλίου και έχετε λάβει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα ε, αποτελέσματά τους και τα έχουμε και στα έγγραφα της ε, συνεδρίασης. Παρακαλώ να τα ελέγξετε. Σημείο τρίτο, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 19ης Ιουλίου και 11η και 12 η Ιουλίου. Μάλιστα. Εγκρίθηκαν τα πρακτικά. Τέταρτο σημείο. Δεν έχουμε ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες δύο οργανικές διαπραγματεύσεις στη σημερινή μας συνεδρίαση. Και περνάμε μέσα στο σημείο 5, προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Θα δώσω το λόγο στο συντάκτη του νομοδότης, τον κύριο Σιλικιώτη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ήθελα να καλωσορίσω όλους τους συναδελφούς στη, μετά τις διακοπές σε μια, στην τελευταία μας χρονιά και ελπίζω αυτή η χρονιά να είναι παραγωγική για την Επιτροπή μας. Ε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδελφούς για την επιδοκομοδητική συνεργασία και τις τροποποιολογίες που έχουν καταθέσει. Ήδη επεξεργαζόμαστε συμβαστικές τροπολογίες ε, για τις συναντήσεις που θα έχουμε προσεχώς με τους κοιόδης ηγητής βάση της γνωμοδότησή μας ε, για τους Western Employers είχαμε θέσει έξι αρχές. Η πρώτη αρχή είναι τη διεύρυνση της οδηγίας και σε εργασιακούς δόμους. Το δεύτερο, τη διεύρυνση του ορισμού του ποιο μπορεί να ονομάσεται Western Employer, αν είναι μόνο εργαζόμενο σε εταιρεία ή αν μπορεί να είναι δημοσιογράφος ή μέλος της οικογένειας. Το τρίτο είναι τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού προστασίας των Western Employers το τέταρτο, την κατάργηση τη υποχρεωτική ιεραρχία καταγγελία, δηλαδή να μπορεί κάποιο να καταγγέλει και κατευθείαν στι αρμόδιε αρχέ ή τα μέσα μαζική επικοινωνία. Πέπτον, τη διασφάλιση τη ανωνυμία ε, του whistleblower, εάν αυτό ή αυτή το επιθυμεί. Και τελευταίο, το έκτον, τη διεύρυνση τη οδηγία και για δημόσιου και ημιδημόσιου οργανισμού. Μέσα από τι δικέ μα τροπολογίε προσπαθήσαμε να ενδυναμώσουμε αυτέ τι θέσει αλλά και να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα που υπήρξαν, όπω για παράδειγμα η διεύρυνση τη ισχύω τη οδηγία μέσα από το παράρτημα 1 και 2. Στι τροπολογίε που κατατέθηκαν υπάρχει γενικά μια σύμπλευση σε αρκετά θέματα. Τέτοια θέματα είναι η προστασία και η δημιουργία εμπιστοσύνη για του whistleblowers, η κάλυψη και εργασιακό θεμάτων στην ισχύ τη οδηγία, αλλά και η διεύρυνση οδηγία για ε, δημόσιου και μη δημόσιου οργανισμού. Προκλήσεις ίσως να υπάρχουν και ε, διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με το άρθρο 13 και πώς ε, διαχειριζόμαστε την ενεργεία στους τρόπους που γίνεται μια καταγγελία αλλά και στον ορισμό του whistleblower. Ε, εμείς όσοι εισηγητής θα προσεγγίσουμε το θέμα με ένα ανοιχτό πνεύμα και ελπίζω να βρούμε λύσει στι δύο συναντήσει των σκιωδών εισηγητών και των βοηθών που θα έχουμε στο επόμενο ε, χρονικό διάστημα. Ε, θα ε, λάβουν οι σκιώδει εισηγητέ στι συμβαστικέ προλογίε εν ευθέτω χρόνο και αναμένω σε περαιτέρω συνεργασία με του σκιώδει εισηγητέ και με όλα τα μέλη τη Επιτροπή ώστε να ολοκληρώσουμε αυτή την γνωμοδότηση ε, με τον καλύτερο τρόπο, με μια συλλογική προσπάθεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιλικιώτη. Θα δώσω το λόγο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τον εκπρόσωπό του που είναι ο κύριος Μπέκερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε στα αγγλικά ο κύριος Μπέκερ. Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος του κυρίου Κάζα που είναι σκιώδης ηγητής, έχει άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις και απουσιάζει. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη δική του θέση. Πρώτον, πολλές ευχαριστίες ε, στον κύριο Σιλικιώτη για το έργο του στο σχέδιο της νομοδότησης. Ε, στη δική μου παρέμβαση θα αναφέρω μερικά σημεία Στι τροπολογίε τα λέω πιο λεπτομεριακά. Γενικά θα ήθελα να αναφέρω ότι ε, είμαστε ικανοποιημένοι από το έργο του εισηγητού σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν πολλές θετικέ τροπολογίε που έχουν προτείνει και άλλοι συνάδελφοι. Επίσης έχω κάνει και εγώ πολλές τροπολογίε που θεωρώ ότι βελτιώνουν το κείμενο. Έχω κάνει πολλές προτάσεις που έχουν στόχο να ε, διαγραφούν ε, κάποιες ε, επαναλήψεις που βαραίνουν το κείμενο, κάποιοι κατάλογοι ας πούμε που κινδυνεύουν να κρύψουν άλλα στοιχεία πιο σημαντικά που θα έπρεπε να καλύπτει αυτή η οδηγία. Οι προτάσεις αυτές καλύπτονται από τις τροπολογίες 69, 71 και 91. Πρέπει να πω ότι από προσωπική εμπειρία που έχω και από την εργασία μου σε αυτό το τομέα και ως εισηγητής, αλλά και από άμεση επαφή που έχω με whistleblowers, πιστεύω ότι η οδηγία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει επιπλέον ασφαλιστικές δικλίδες και να φροντίζει να προστατεύει τους καταγγέλλοντες αυτούς όταν εκθέτουν ε, υψηλά ιστάμενα πρόσωπα και κυβερνητικά στελέχη. Παίζουν σημαντικό ρόλο οι καταγγέλλοντες για να προλαμβάνονται οι καταχρήσεις και η διαφθορά και θα πρέπει να θεωρούνται ένας μηχανισμός λογοδοσίας που να υπάρχει έτσι ε, έλεγχος δημόσιος των κυβερνήσεων. Είναι σημαντικό τα πρόσωπα αυτά να χαίρουν ε, επαρκούς προστασίας και κατάλληλες. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να αναφέρουν ε, στη δικαιοσύνη ε, στα κράτη-μέλη ε, απευθείας και να λαμβάνουν προστασία. χωρίς να εξαρτώνται από εκείνους τους οποίους κατηγορούν και για τους οποίους έχουν επιβαρυντικά στοιχεία. όταν φέρουν πληροφορίες, ε, όταν αποκαλύπτουν πληροφορίες. Προσβλέπω στη στενή συνεργασία με τον εισηγητή και τους κοιόδες εισηγητές τις επόμενες ημέρες για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη γνωμοδότηση αυτή και να υποστηρίζουμε ε, τους ε, καταγγέλλοντες που αναφέρουν παραβιάσεις ή καταχρήσεις στο ενωσιακό δίκαιο. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική μέχρι τώρα συνεργασία μας. Η πρόεδρος ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Τέτσιν. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ε, κοίταξα και εγώ τις τροπολογίες και ε, χαίρομαι που συμφωνούν στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και άλλες πολιτικές ομάδες, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της περιορίζεται σε κάποιους τομείς και μόνο του ενωσιακού δικαίου. Πιστεύω ότι ο προσανατολισμός ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η προστασία της εσωτερικής αγοράς. Εγώ θέλω να διευρυνθεί και στο εργατικό δίκαιο και στις εργασιακές συνθήκες και στα δικαιώματα των συνδικαλιστών και εκπροσώπων των εργαζομένων. Κατά τα άλλα, έχω διευρύνει και τον κύκλο προσώπων. Μεταξύ αυτών και πρόσωπα που δεν είναι στις κλασικές μορφές απασχόλησης και εργασίας και τα μέλη των οικογενειών τους που θα πρέπει να ενταχθούν στην οδηγία. Αυτό είναι και θέση της ε, έκθεσης πρωτοβουλίας Επιτροπής μας πέρυσι. Επίσης, σημασία για μένα έχει το σημείο της συνέχειας που δίνεται στην καταγγελία. Έχουμε και αντίστοιχες νομολογίες και θα πρέπει να κινηθούμε με βάση αυτές. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει μια συνέχεια πρώτα εσωτερική και μετά εξωτερική και σωστό είναι αυτό. Διαρωτώ με όμως τι συμβαίνει. Όντως έχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίω για τους καταγγέλλοντες, τους whistleblowers, αρκεί και μόνο να ακολουθήσουμε την ομολογία που ήδη υπάρχει. Θα το ξανασυζητήσουμε στον κύκλο των σκιωδών ε, εισηγητών και θα πούμε και τα υπόλοιπα και τις λεπτομέρειες. Πώς θα το ε, ρυθμίσουμε ακριβώς στο κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Uh, ε, Mr. Hodge is not here. Ο κ. Hodge δεν είναι εδώ. κύριε Μάκεντάρ, τον εκπροσωπεί. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κ. Χότς λυπάται, δεν μπορεί να παραστεί σήμερα μου ζήτησε να σας παρουσιάσω τη θέση του. Θέλω να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Έχει δύο τροπολογίες, έχει υποβάλει δύο τροπολογίες εκ μέρους του ECR. Πρώτον για το άρθρο 1. Πιστεύει ότι ε, ο κλειστός κατάλογος θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ανοιχτό κατάλογο που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα όσα αναφέρει η οδηγία και τα κράτη-μέλη να μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα όρια στην εθνική του νομοθεσία. Ο κατάλογος περιλαμβάνει πιο σημαντικές, ε, πιο σημαντικούς τομείς, αλλά ορισμένα κράτη-μέλη μπορούν να θέλουν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογή για να προστατεύσουν του μάρτυρε δημοσίου συμφέροντο και για θέματα τα οποία δεν αναφέρονται στην πρόταση. Μια τέτοιου είδου διεύρυνση δεν θα επηρεάζει την προστασία στις, στους τομείς οι οποίοι ήδη αναφέρονται, ενώ θα διεύρυνε το πεδίο εφαρμογή των ατόμων τα οποία μπορούν να λάβουν το χαρακτηρισμό του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα αυτό και με την αιτιολική έκθεση. Σύμφωνα με την παρούσα πρόταση, η διεύρυνση της προστασίας σε άλλους δεν απαγορεύεται, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποτελούσε και εφαρμογή της οδηγίας. Θα ήταν πιο χρήσιμο αν η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος ήταν ίδια για όλους ανεξαρτήτως του τομέα με βάση τον οποίο ε, καταγγέλουν. Δεύτερη τροπολογία αφορά το άρθρο 2 παράγραφος 1.c. Ο κ. Χότς θεωρεί ότι η διεύρυνση της προστασίας τους εθελοντές είναι υπερβολική και ότι η προστασία θα πρέπει να αφορά μόνο ατόμα τα οποία επηρεάζονται άμεσα οικονομικά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία. Πρόεδρος. Κυρία Τούμ, από τους φιλελεύθερους είναι εδώ, δεν είναι εδώ, όχι. Υπάρχει κάποιος άλλος που να εκπροσωπεί τους φιλελεύθερους. Όχι. Κύριος Λάμπαρτ, για τους Πράσινος. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Ε, πολύ καλή συνεργασία ως τώρα και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Συμφωνούμε με κάποια από τα πόσα είπαν οι προηγούμενοι. Σε ό,τι αφορά τους τομείς που καλύπτονται, Ήδη κάποιοι ζήτησαν να, να διευρυνθούν και στο ε, εργασιακό δίκαιο και εμείς έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες, ιδιαίτερα στην ετωλική έκθεση, αλλά και στο άρθρο 1 και το σχετικό παράρτημα ε, του τι ακριβώς θα σήμαινε εργασιακό δίκαιο. Όπως και άλλοι συνάδελφοι έχουμε υποβάλει τροπολογίες σε ό,τι αφορά την ανωνυμία του καταγγέλλοντος. Πολλές ε, φορές η αποκάλυψη της ε, ταυτότητας του μάρτυρα έχει οδηγήσει σε σημαντικό πλήγμα για τον καταγγέλλοντα. Θα πρέπει να προστατεύεται. Η προστασία επίσης είναι σημαντική ανεξαρτήτως της ισορροπίας δυνάμεων στο εργασιακό περιβάλλον. Ακόμα και εκεί που έχουμε οριζόντια σχεδόν ε, διοίκηση, ε, ακόμα και εκεί υπάρχει μια συγκεκριμένη ισορροπία δυνάμεων και εξουσιών που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης κάποιοι είπαν για την συνέχεια που δίδεται στις καταγγελίες έτσι ώστε να ενημερώνεται ο καταγγέλων, να είναι ενήμερος της προόδου και των πορισμάτων. Επίση θέλουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή για να συμπεριληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ε, σχετικές ε, οργανώσεις. Υπάρχει επίσης και ένα θέμα σε ό,τι αφορά τις, ε, την ιεραρχία των εκθέσεων. Δεν είναι σαφής. Πρέπει επίσης να ενισχυθεί η προστασία του καταγγέλλοντος. Το έχουμε εξετάσει και στο παρελθόν, γνωρίζουμε πολύ καλά τα θέματα τα οποία εμφανίζουν τα προβλήματα. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, μέτρα, ε, αντίμετρα τα οποία μπορεί να ληφθούν ε, τιμωρητικά ή εκδικητικά από πλευράς των καταγγελωμένων. Ευχαριστούμε πολύ τους και και τον εισηγητή. Ε, κάνουμε πολύ καλή δουλειά και ελπίζουμε ότι το τελικό κείμενο θα είναι πολύ ισχυρό. πολύ μεταξύ αυτών εμείς η ομάδα μου, το επιθυμούμε εδώ και πολύ καιρό. Ευχαριστούμε. Ο δεν εκπροσωπεί εδώ πέρα το EFTD από όσο βλέπω. Άρα το ENF τώρα έχει το λόγο. Κύριε Μαχτάν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. κυρία Μόλεκεμ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG Just ενδεχομένω βρίσκεται στην αίθουσα. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κατέγραψα όλες τις παρατηρήσεις Διάβασα μάλιστα και τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για τη γνωμοδότηση αυτή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Ενδεχομένως θα μπορούσα να επιμείνω περισσότερο σε ένα σημείο που έχει να κάνει με την συμπερίληψη του εργασιακού δικαίου. Ενδεχομένως εδώ πέρα να προκύψει ένα ζήτημα με την νομική βάση, αν κάνουμε κάτι τέτοιο. Ξέρετε ότι η νομική βάση προβλέπει ότι η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους πριν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε αυτό πρωτού υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της σε αυτή την φάση, καθότι δεν κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθεί το εργασιακό δίκαιο, δεν είμαι σίγουρη ότι θα είναι δυνατό να συμπεριληφθεί μετά την επίσημη υποβολή της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκ των υστέρων δηλαδή, γιατί μπορεί να εκλειφθεί ως παράκαμψη της επίσημης διαδικασίας, ακριβώς επειδή επί του σημείου αυτού δεν έχει γίνει πρώτερη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Ενδεχομένως να πρέπει να σας απασχολήσει λίγο περισσότερο το σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ξαναδώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σελικιώτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι αρκετά σύντομο. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για τα καλά του λόγια και για την επικοδομητική ε, συνεργασία. Ε, είπα και στην αρχική μου εισήγηση ότι οι τροπολογίε βελτιώνουν το κείμενο ε, και ε, υπάρχουν κάποια ζητήματα που ω θέματα αρχή τα παρέθεσα στην αρχική μου παρέμβαση, τα οποία πρέπει βεβαίω να επιμένουμε. Ε, στόχος μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι πρώτα-πρώτα να υπάρξει προστασία των καταγγέλλοντων, των whistleblowers, ε, ε, να μπορεί να διατηρείται η, η, ανωνυμία, ε, να δημιουργηθεί βέβαιος και μέσα από αυτή τη διαδικασία ένας μηχανισμός λογοδοσίας των δημόσιων προσώπων. Συμφωνώ που τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν να υπάρξει ε, και ε, ε, ανωνυμία ώστε να μπορούν να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία για τους καταγγέλλοντες και βεβαίως να υπάρξει η ενημέρωση. Έχουμε πει και άλλες φορές στο παρελθόν ότι η διαφάνεια ποτέ δεν βλάπτει. Αντίθετα, βοηθά ακριβώς να ασκείται καλύτερα η εξουσία και να περιορίζονται φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Ε, ήθελα να ολοκληρώσω κάνοντα ένα ε, ε, σχόλιο σε αυτό που είπε και η εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιλαμβάνομαι αυτό που είπε για την νομική βάση, όμω εμεί ω Κοινοβούλιο είμαστε υπόχρεοι να θέτουμε αυτό το ζήτημα και πρέπει να το θέσουμε. Εδώ υπάρχει, θα έλεγα, μια ε, καθολική συμφωνία ότι πρέπει να επεκταθεί και στο εργασιακό δίκαιο. Και εδώ είμαστε ακριβώ να βρούμε του τρόπου για να επεκταθεί και στο εργασιακό δίκαιο και να καλύψει μάλιστα όπως είπαν και άλλοι συναδέλφοι και ομάδες που δεν καλύπτονται ε, μέσα από τα ε, επαγγέλματα ε, γιατί ο στόχος μας είναι, επαναλαμβάνω, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία για τους καταγγέλλοντες, για τους whistleblowers. Και εδώ είναι που εμείς πρέπει να, το, να επιμένουμε σε αυτή τη θέση για την επέκταση στο εργασιακό δίκαιο και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα θεσμικά όργανα βρουν τρόπους για να μπορεί αυτό να καταγραφεί και στην οδηγία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιλικιώτη. Στην Επιτροπή Απασχόλησης θα ψηφίσουμε στις 24 Σεπτεμβρίου και στη Γιούρη θα ψηφίσουμε στις 10 Οκτωβρίου. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία μας, σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Ας περιμένουμε όμως δύο λεπτά. Πρωτού ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, μπορούμε να κάνουμε και μία δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε πόσοι είμαστε και ενδεχομένω να καταφθάσουν και περισσότερα μέλη στην Επιτροπή. Okay, friends, then we... Αγαπητοί φίλοι, ας ξεκινήσουμε την ψηφοφορία μας. Καταρχάς θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019. Συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική παλήθευση για τη συμβαστική Α. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εκρίνεται 31 υπέρ 10 κατά. Περνάμε στη βαστική Β, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία. Συγγνώμη. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 13, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 35 κατά 8 υπέρ. Περνάμε σημαστική D. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική E υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9, τροπολογία 26 τώρα υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία H. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίσουμε τώρα το σχέδιο γνωμοδότησης ε, όπως τροποποιήθηκε. Μονομαστική κλίση. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται 32 υπέρ, 10 κατά και μία αποχή. να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια, την υποφαινόμενη δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ για την... Ε, να ευχαριστήσω μάλιστα και το προσωπικό μας για την όλη υποστήριξή τους, οι οποίοι εργάστηκαν μάλιστα κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Ας περάσουμε τώρα στις τροπολογίες επί του προπολογισμού. Employment 5500 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5501 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για το 5501. Άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 24 κατά 18 υπέρ. 55-02 τώρα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλα 55-03 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εμπλα. 55 55-04 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλα 5505 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 5506 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 5507 τώρα υπέρ παρακαλώ. Α, μάλλον δεν την ψηφίζουμε αυτήν. Όχι, πρέπει να την ψηφίσουμε τελικά. Υπέρ παρακαλώ της 5507. Έχει γίνει λάθος, έχει γίνει λάθος στον κατάλογο σας που λέει no vote. Πρέπει παρόλα αυτά να ψηφίσουμε την 5507. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλει ηλεκτρονική επαλήθευση. Πολύ ωραία. Ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την 5507 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Κυρία Σίπελ, ζητεί το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο όμως. Χωρίς μικρόφωνο. Καλά και με ισοψηφία απορρίπτεται όμως. Ε, έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ψήφια. So, um, it's 21, 22. Mm, it's 21, 22. Uh, Το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδατε. 22 κατά 21 υπέρ, άρα απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την έμπλη 5508. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5509 καταπίπτει και περνάμε έτσι στην έμπλε 5510. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5511 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλε 5512 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλ 5513, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλ 5514, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλ 5515, υπέρ παρακαλώ. Α, με συγχωρείτε, καταπίπτει λέει πρόεδρος. Περνάμε έτσι στην έμπλη 5516 υπέρ, κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 5516 άρχιτη ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται. Ισοψηφία 23 υπέρ, 23 κατά. Άρα απορρίπτεται. Έμπλ 55-17 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 55-19 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55.20 υπέρ. Ακαταπίπτει αυτή. Περνάμε έτσι στην ΕΜΠΛ 5521 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. ΕΜΠΛ 5543 αποκινούμε την 5544 είναι ταυτόσιμες υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνονται. ΕΜΠΛ 5524 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. ΕΜΠΛ 5525 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε ονομαστική κλίση τώρα τώρα την 5526. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 υπέρ, 21 κατά και μία αποχή. Έμπλε. 55-27 τώρα, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλε 55-28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλε 55-29 υπέρ, κατά, αποχές. Ας ε, ελέγξουμε την 55-29 ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Σας πεθυμίζω ότι ψηφίζουμε την 5529 29 πέρας και απορρίπτεται. 43 κατα εμπλ 5530 τώρα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία λοιπόν. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. 20 υπέρ 26 κατά. Έμπλ 55-31 υπέρ κατά αποχές. Ας ε, ελέγξουμε ηλεκτρονικά και για αυτήν. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 45 υπέρ, 1 κατά. Ε, μάλλον πρέπει να συνέλθω λίγο να ξεκουραστώ από τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Έμπλ 55-32 υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές, μάλλον να απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την 5532, άρτη ψηφοφορία, πέρας. Και όντως απορρίπτεται. Περνάμε έτσι στην έμπλε 5533. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές Ας την ελέγξουμε και αυτήν ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο Περνάμε στην έμπλ 5534. Τώρα αποκινούμε την έμπλ 5535. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Έμπλ 5536. Υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά και την 5536 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. 27 υπέρ. Εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε στην έμπλα 5537 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, έμπλη 5538 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, έμπλη 5539 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, έμπλη 5540 υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται, έμπλη 5541 υπέρ, κατά Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 5541 άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. Έμπλη 5542 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν προβλέπεται τελική ψηφοφορία για τις τροπολογίες αυτές. Ολοκληρώσαμε λοιπόν. Ολοκληρώσαμε για σήμερα για την ψηφοφορία τουλάχιστον ολοκληρώσαμε. Προφανώ εκκρεμούν ακόμα κάποια σημεία στη μερίσια διάταξη σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σα, λέει πρόεδρο, και θα συνεχίσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο συζητήσαμε και στο παρελθόν, στην τελευταία συνεδρίασή μας, αν δεν κάνω λάθος, πριν τις θερινές διακοπές, κάναμε μία εις συζήτηση όσον αφορά την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Θα εξετάσουμε σήμερα, την εξέταση, θα εξετάσουμε σήμερα τις 975 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για την πρόταση αυτή κανονισμού που θεσπίζει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Λένερς, ο οποίος θα μας κάνει μια εισαγωγική παρέμβαση και θα δώσω εν συνεχεία το λόγο στους κοιόδης συγητές. Κύριε Λένερς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, έχει ήδη γίνει μια πολύ ειλικρινή συζήτηση για αυτό το θέμα, συγκεκριμένα στις 11 Ιουλίου, πριν διακόψουμε για το καλοκαίρι. Οι συνάλφοι στήριξαν με θέρμη το σχέδιο έκθεσης Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας περάσαμε πολλές ευχάριστες ώρες κατά τη διάρκεια των καθερινών μας διακοπών δίπλα στη θάλασσα ή στην πισίνα εξετάζοντας τις τροπολογίες. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά οι συνάλφοι στο παρελθόν έδειξαν ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό το θέμα, το έχουν στην καρδιά τους 929 ήταν οι αρχικέ τροπολογίε μαζί με τις δικές μου 975. Αυτός ο αριθμός δείχνει ότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είπα και τον Ιούλιο. Είναι το κομμάτι που λείπει από το puzzle σε ό,τι αφορά την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα και τον Ιούλιο, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε σαφείς, αυστηρούς και εφαρμόσιμου κανόνε σε ευρωπαϊκό πέδο σε ό,τι αφορά την κινητικότητα του ορατικού δυναμικού. Ήδη έχουμε την ε, πλατφόρμα των, της αντίλωτης έχουμε την ε, οδηγία απόσπασης και άλλες προτάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή συζητώνται. Χρειάζεται όμως και καλύτερη εφαρμογή. Ιδιαίτερα διασυνοριακή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων κινητικότητας. Οι Ευρωπαίοι γίνονται όλο και πιο κινητικοί. 17 εκατομμύρια πολίτε εργάζονται ή ζουν σε κράτη-μέλη εκτό του δικού τους. Οπότε θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διασυνοριακή διάσταση της εφαρμογής των κανόνων. Πρότεινα αυτή η αρχή να έχει περιορισμένο πεδίο και να εστιάζει στην εφαρμογή, προκειμένου να κάνει τη διαφορά. Δεν έχει νόημα να δημιουργήσουμε ένα μαστόδοντα, μια αρχή με πολύ ευρία εντολή που δεν θα μπορεί να δράσει. Αυτά τα είπα και τον Ιούλιο. Τώρα για τις τροπολογίες. Θυμήθηκα το Ρωμαίο και την Ιουλίατα στην αρχή, γιατί πολλοί συνάλφοι ανέφεραν, ζήτησαν να αλλάξει το όνομα, να την ονομάσουμε ε, αρχή κινητικότητας των εργαζομένων, ευρωπαϊκή αρχή, συνοριακά θέματα της ε, ε, αγοράς, κάτι που δίνει αρχικά πολύ περίπλοκα Ελπίζω να μην χρειαστεί να φορτώσουμε με τέτοιου είδου όνομα την αρχή αυτή. Πάντως είναι πιο σημαντικά τα καθήκοντα και η αποστολή ε, της αρχής αυτής από ότι το όνομα. Ελπίζω θα βρούμε μια λύση για το όνομα που θα αντικατοπτρίζει και τα καθήκοντα τα οποία θα τη ανατεθούν. Θέλω η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας να εστιάζει στην εφαρμογή. Και οι περισσότεροι συνάδελφοι πραγματικά συμφωνούν προσπαθώντας να περιορίσουν τα καθήκοντα της αρχής για να είναι πιο αποτελεσματικοί. Κάποιοι συνάδελφοι ε, ζήτησαν να διαγραφούν τα περισσότερα από τα καθήκοντα επίσης. Νομίζω ότι αυτό θα καθιστούσε την αρχή υπερβολικά συγκεντρωμένη σε πολύ λίγα πράγματα. Θέλουμε να είναι και αποτελεσματική. Πάντως, ένα μεγάλος αριθμός συναδέλφων είναι ε, υπέρ ε, του περιορισμένου, του περιορισμού του, των ενημερωτικών καθηκόντων της ε, αρχής, όπως προτείνω εγώ. Επίσης υπάρχουν κάποιες διαφορές σε ό,τι αφορά την παράγραφο που διευκολύνει τη συνεργασία ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους σε περιπτώσεις διατάραξης των ουσιακών σχέσεων διασυνοριακά. Είναι φυσικό καθήκον της αρχής και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη τις ερχόμενες εβδομάδες. Επίσης θα μπορούσε να διευκολύνει κοινέ ή συντονισμένε επιθεωρήσεις. Σε αυτό οι γνώμες διχάζονται. Δεν είναι σίγουροι οι συνάδελφοι ούτε για την ανάγκη τέτοιων επιθεωρήσεων, ούτε και για το κατά πόσον οι Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα πρέπει να διευκολύνει να συμμετέχει σε τέτοιου είδου ελέγχου. Και επίσης δεν ξέρουμε αν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να είναι υποχρεωτικό ή εθελοντικό. Έχουμε λοιπόν θέματα να συζητούμε με τους κοιόδης ηγητές για αυτό το ζήτημα. Είναι από τα σημεία κλειδιά όμως πρόταση. Ελπίζω ότι θα βρούμε μια ικανοποιητική λύση. Τώρα, υπάρχουν και κάποιες ασάφειες στις τροπολογίες. Για παράδειγμα, πολλές ε, τροπολογίες για καινούριου ορισμούς. Η πρόταση είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας να ασχολείται μόνο με κανόνες που ήδη υφίστανται και έχουν ορισμό. Καλό θα ήταν λοιπόν να αποφύγουμε την, να δώσουμε καινούριου ορισμούς σε αυτή την πρόταση. Άλλα θέματα, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ορισμένε διαδικασίες. ο ρόλος της Διοικητικής, της ε, Διοικητικής Επιτροπής, η, ο ρόλος της ε, αρχής στην διερεύνηση παραβιάσεων των, της ε, νομοθεσία. νομοθεσίας, η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών δεν είναι εύκολο να τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα. Θα το κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες με τους κοιόδης εισηγητές και όλους όσοι ενδιαφέρονται. Ο στόχος μου σε αυτήν την έκθεση ήταν να εξασφαλίσω την ισορροπία ανάμεσα στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και την επικορικότητα αφενός και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια πραγματική αρχή που θα εφαρμόζει αποτελεσματικά τους κανόνες της αφετέρου. Ελπίζω αυτή την ισορροπία να τη διατηρήσουμε και στο τελικό κείμενο όταν το ψηφίσουμε. Και ελπίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα. Μια ακόμα φορά ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους και ελπίζω θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Λέναρς. Σκιώδης πρώτα και μετά τα υπόλοιπα μέλη που ζήτησαν το λόγο. Ο κύριος Πυρίνσκι πρώτος, σοσιαλιστής και δημοκράτης, σκιώδης ηγητής. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, and... Uh, Χαίρομαι που σας ε, ξαναδέλφω. Ξαναβλέπω και τον κύριο Λένας και τους συναδέλφους για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό και γεμάτο προκλήσεις Μα σου και η έκθεση. Όπως είπε ο κύριο Λένας, 975 είναι τροπολογίες. Καταλαβαίνετε, αυτό μιλάει από μόνο του και δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Θα ήθελα επίση να πω το εξή. Η δική μας γενική προσέγγιση στις τροπολογίες ποια είναι θέλουμε να προσπαθήσουμε να τα βρούμε σε μια ε, ισόρροπη προσέγγιση, όπως είπε και ο ίδιος ο εισηγητής, να δημιουργήσουμε ένα θεσμό, μια αρχή που έχει πραγματική προστιθέμενη αξία. Και να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά εργασίας ε, στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Και υπό την έννοια αυτή κύρια Πρόεδρε. Για μας έχει σημασία να προσπαθήσουμε να ορίσουμε με τρόπο και όρους πιο συγκεκριμένους τι είναι αυτή η ισορροπία και ποια είναι η ισόρροπη προσέγγιση και πώς θα φτάσουμε στην ισορροπία αυτή. Τρεις είναι λοιπόν οι τομείς που έχουν γενικά σημασία και θέλω πραγματικά να τους έχουμε υπόψη μας. Το πρώτο είναι βεβαίω οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογή και το πεδίο δραστηριοτήτων της αρχής. Δεύτερο, τα καθήκοντά της ε, και πώς θα τα ορίσουμε για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Και τρίτον, οι δομές. Αρχίζω λοιπόν από του στόχους. Ω σοσιαλιστέ και δημοκράτε καταθέσαμε περίπου 125 τροπολογίε. Ε, με μονομένες συνάδελφοι μαζί με άλλους έχουν κάνει τροπολογίες και όλα αυτά αντανακλούν την επιθυμία μας να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας όσο γίνεται πιο αποτελεσματική. Ένα σημείο αρχής, κυρία Πρόεδρε, προσπαθήσαμε να βασίσουμε την προσέγγισή μας στο κείμενο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αιτιολογική Σκέψη 1. Δηλαδή, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η ελεύθερη εγκατάσταση και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών είναι θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατοχυρώνονται δε και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχουν αυτές οι τρεις ελευθερίες οι οποίες Ε, έχουν να κάνουν με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που αναζητούν εργασία και θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, εφαρμόζονται σωστά αυτές οι τρεις ελευθερίες οι οποίες συνδέονται και μεταξύ τους. Και να αναφέρω εδώ μια πολύ συγκεκριμένη τροπολογία που θεωρώ απαράδεκτη. Είναι η τροπολογία 54 που προσθέτει στο κείμενο ε, του, της σκέψης το εξής. Τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας, ωστόσο, δεν είναι απόλυτα. Και θα πρέπει να αποτρέπεται καταχρηστική ε, κατάχρηση μάλλον αυτών των ε, ελευθεριών. Αυτό μπορεί να εμφανιστεί και στα τρία και έχουμε δει δραστική ε, κατάχρηση μέχρι και εγκληματική ε, κατάχρηση από διάφορες εταιρείες, θηρίδες, μαϊμούδες κλπ. Πολύ σοβαρά και εγκληματικά φαινόμενα στην παροχή υπηρεσιών. Αυτό δεν είναι ισορροπία και δεν συμφωνώ με τέτοιες προτάσεις και προσεγγίσεις. κατανοούμε το στόχο που ανέφερε και ο κύριος Λέναρτς να εφαρμόζεται με σωστό τρόπο το κείμενο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλά να επικεντρωθούμε μόνο στην ε, ε, εφαρμογή του νόμου και στην επιβολή του νόμου και να είναι αυτός ο φάρος μας, ε, πολύ μονομερές. Θα πρέπει να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα, ποια είναι τα αίτια των προβλημάτων, να προσπαθήσουμε να τα καταργήσουμε. Υπάρχουν διάφορες διακρίσεις που βασίζονται σε διάφορες αδικίες και ανισότητες που δημιούργησε η αγορά όταν αφήθηκε ασίδωτη. Από την άλλη λοιπόν να γίνει μια σωστή ανάλυση του κινδύνου, της συνεργασίας με ανταλλαγή ε, πληροφοριών, με εξέταση των αιτίων, επαναλαμβάνω, των διαφόρων στρεβλών, καταστάσεων και καταχρήσεων σε περίπτωση που παρατηρούνται στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Οπότε, επαναλαμβάνω ότι για την ομάδα μας το πρόβλημα δεν είναι μόνο ε, στην απόσπαση των εργαζομένων και παραβιάσει του κοινωτικού δικαίου, αλλά και ε, όταν ε, μετακινούνται οι εργαζόμενοι για να κατασταθούν σε ένα κράτος μέλος και στην αγορά εργασίας. Και στο τέλος ανέφερε κάτι ο κύριος Λέναρτ σχετικά με τους ορισμούς. Είναι γεγονός ότι Υπάρχουν διάφορα νομοθετήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιλαμβάνουν ορισμούς, αλλά κατά τη διάρκεια της σύνταξης των τροπολογιών διαπιστώσαμε αποκλήσεις ε, στους ορισμούς για την ίδια δραστηριότητα. Διαφωνώ λοιπόν με τον κύριο Λέναρτ, Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε και νέους ορισμούς. Αυτό θα βοηθήσει ε, το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας ε, και δεν θα την παρεμποδίσει πόσο δε περισσότερο που σήμερα δεν έχουμε κοινή αντίληψη για τον ορισμό του εργαζομένου. Τι εστί εργαζόμενος, επειδή αλλάζει η φύση της εργασίας. Και αν ε, ε, ο οργανισμός, ε, η αρχή αυτή θέλουμε να έχει ρόλο πρωταγωνιστικό και σημαντικό, πρέπει να καταλάβουμε γιατί πράγμα μιλάμε ποια είναι η δραστηριότητα και ποιο είναι ο εργαζόμενος ή αυτός που ασκεί τη δραστηριότητα αυτή. Είμαι ακόμα στο πεδίο εφαρμογή, κυρία Πρόεδρε. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπόψη κάποιες πρακτικές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, γιατί φοβούνται ότι θα διαταραχθεί ένα σύστημα που λειτουργεί σωστά. Υπάρχει η περίφημη ρήτρα Μόντι που λαμβάνει υπόψη της αυτές τις ανησυχίες και απαντά σε αυτές και θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο κείμενο. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες για τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Αρχής γιατί δεν έχουμε τόσο χρόνο. Είναι πραγματικά, είπαμε, τεράστιος όγκος των τροπολογιών. Αλλά όταν συζητούμε για ανταλλαγή προφοριών, συνεργασία, ε, κοινέ επιθεωρήσεις, διαμεσολάβηση, επίλυση διαφορών κτλ. Η βασική μας ε, πηξίδα εκεί θα πρέπει να είναι η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Αρχή Εργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Σε καμία περίπτωση η σχέση αυτή δεν θα πρέπει να είναι κάθετη. Ε, υπάρχει μια συνεργασία η οποία θα οικοδομηθεί με σεβασμό πάντα στις αρμοδιότητες και εξουσίες των κρατικών αρχών αλλά να έχει και ένα ε, ακέραιο ρόλο η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας στο συντονισμό ε, των εθνικών αρχών και στο να τις κάνει να καταλάβουν τι σημαίνει η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Και από εκεί και πέρα να τις βοηθάει και όλες να ξεπερνούν κάποιες δυσκολίες και να λύνουν κάποιες διαφορές. Για τις δομές τώρα που είναι το τρίτο, τηλεγραφικά κυρία Πρόεδρε, εμείς δεν πιστεύουμε ότι είναι καλή ιδέα να ενταχθούν οι δομές ε, του συστήματος EURES στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Καλά δουλεύει και λειτουργεί, γιατί να το πειράξουμε το σύστημα EURES. Ε, είδαμε κάποιες τροπολογίες που φιλοδοξούν στην αλλαγή του καθεστώτος που τελείωσε έληξε το 2016, αλλά εμείς δεν πιστεύουμε ότι στην οδηγία αυτή θα πρέπει να ε, καλυφθούν τα ζητήματα του με τροπολογίες κλπ. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Το ίδιο ισχύει και για την Διοικητική Επιτροπή για την Κοινωνική Ασφάλεια και η ιδέα που εκφράστηκε να μεταβιβαστούν κάποιες αρμοδιότητες, να χωριθούν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Επασχόλησης Εργασίας δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Ούτε συμφωνούμε με την ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαλυθεί μια άλλη πλατφόρμα να μην διακοπεί μια διαδικασία για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Και τέλος, υπάρχει και μια ανάγκη που αισθανόμαστε πάρα πολύ έντονοι να υπάρχει μια τριμερής μορφή ε, στην ΕΛΑ και να υπάρχει και ένα εκτελεστικό όργανο, διοικητικό συμβούλιο, για να ε, λειτουργεί καλύτερα. Και σε ό,τι αφορά το όνομα, συμφωνώ με τον κύριο Λένα που εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με την προσθήκη νέων ε, αρχικών. Να μην γίνει οργανισμός, να παραμείνει αρχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ διευκρινιστικά τα σχόλιά σας για όλους εμάς που δεν έχουμε εμπλακεί στενά στις συζητήσεις. Κυρία Τρεμπίσιος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή μας ε, η πληθώρα των τροπολογιών ε, ήδη αναφέρθηκε και είναι εύγλωτο και αυτό. και έγιναν και διάφορες συγκεκριστικές συζητήσεις για το όνομα. Είναι δύσκολο τώρα να, να παρουσιάσει κανείς όλα αυτά συνοπτικά. Στις δικές μου τροπολογίες που επικεντρώθηκα οι συνθήκες ορίζουν σαφώς ε, τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και τις κατανέμουν σαφώς. Και θέλω αυτό να διαφυλεχθεί και τονίζω ότι ο πυλώνας κοινωνικά δικαιώματα ε, είναι απλώς ε, μια διακήρυξη πολιτικών προθέσεων ή προθέσεων πολιτικής και δεν έχει καμία σχέση με ευρωπαϊκό δίκαιο. Τα κράτη-μέλη ορίζουν πώς οργανώνουν την αγορά εργασία τους και εμείς θα πρέπει να τα συμπληρώσουμε όλα αυτά. Και βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταπολεμάει την απάτη και ε, τις παρανομίες υποστηρικτικά όμως προς τα κράτη-μέλη και πάντα σε συνεννόηση με τις εθνικές αρχές. Κάτι άλλο που έχει μεγάλη σημασία επίσης είναι η ανταλλαγή πληροφοριών για τις διασυνοριακές δραστηριότητες και υποστηρίζουμε να ισχύουν οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς ε, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση. Κάτι άλλο σημαντικό, το είπε και ο συγγετής, οι διπλέ δομέ και επικαλύψεις θα πρέπει να αποφεύγονται. Υπάρχουν ήδη συστήματα που λειτουργούν καλά, όπω είναι το σύστημα Eures. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να εφευρίσκουμε τον τροχό από την αρχή. Επίση, κάτι άλλο που έχει σημασία. Οι εθνικέ αρχέ ε, θα πρέπει όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά να ενταχθούν στην νέα αυτή δομή. Κάτι άλλο που είχα πει και πριν τις νέες διακοπές, προστασία δεδομένων των εργαζομένων σε αυτή τη νέα αρχή και θα χαιρόμουν αν εγκρίνετε τις προτάσεις μου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. Κύριε Χάρκιν για τους φιλελεύθερους. Πρέπει να ομολογήσω ότι αντίθετα με του υπόλοιπου συναδέλφους δεν πέρασα το καλοκαίρι μου διαβάζοντα τι τροπολογίες. Αυτό θα φανεί άλλωστε και από τα σχόλιά μου και, θα, και από τη συντομία τους. Καταρχήν ευχαριστώ τον εισηγητή. Εξετάσαμε ήδη τον Ιούλιο το αρχικό έγγραφο με το οποίο συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσει για θέματα που πρέπει να συζητηθούν κλπ. Είπε ο εισηγητή σήμερα το πρωί ότι δεν έχει νόημα να δημιουργήσουμε έναν ξεδοντιασμένο τίγρη. Η ερώτησή μου είναι, έχουμε νομική βάση για την, στην πρότασή μας, στην πρόταση αυτή για τέτοιου είδους τροπολογίες. Επίσης, λέει ο να περιορίσουμε τον αριθμό των καθηκόντων της αρχής. Για παράδειγμα, πολύ περιορισμένο για καθόλου ρόλο παροχής πληροφοριών. Αν δούμε όμως την έκθεση του ελεγκτικού συνέδριου για την καλύτερη εστίαση της χρηματοδότησης βέβαια, αλλά τότε είχαμε διέξι συστάσεις, εκ των οποίων τρεις αφορούσαν την παροχή πληροφοριών και την ε, συλλογή δεδομένων. Δεν, είμαστε, δεν είμαι εναντίον της κατάργησης αυτής της πτυχής, αλλά Δεν είμαι ε, εναντίον της, ε, της συμπερίληψης αυτού του καθήκοντος, αλλά πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Δεν μπορούμε όμως να το αγνοήσουμε. Επίσης, πολλοί μιλούν για την διασυνοριακή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στον τομέα της εργασιακή κινητικότητα και την αντιμετώπιση των καταχρήσεων. Όπως είπε ο κ. Περίνσκι, η ελευθερία διακίνησης είναι βασική ελευθερία των πολιτών μας, θα πρέπει να διασφαλίζεται, θα πρέπει όμως να δούμε και την αρχή της επικορικότητας. Και εδώ νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, να βρούμε την, το σημείο ισορροπίας ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Γιατί μιλούμε για συνεργασία ανάμεσα σε εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, αλλά πολλές από τις τροπολογίες πηγαίνουν πολύ πιο μακριά ένα από τα θέματα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε είναι η πτυχή της νομικής βάσης για την οποία μίλησα προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά το όνομα, εμένα με ικανοποιεί η πρόταση της Κομισιόν. Αυτά. Τίποτα άλλο προς το παρόν. Κυρία Κάρη. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Με τόσες προτάσεις τροπολογιών δύσκολα θα επιλέξουμε ποιες είναι οι καλύτερες. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αποφασίζοντας ποιος είναι ο στόχος αυτής της αρχής. Για μας ο στόχος είναι να στηρίξει την ενιαία αγορά. όχι να δούμε, όχι προκειμένου να προστατέψει τους πολίτες από το εξωτερικό ντάμπινγκ. Ε, μια καλή αγορά εργασίας, αυτό χρειαζόμαστε. Εμάς μας ενισχύει ιδιαίτερα το θέμα των κοινωνικών εταίρων. Θα πρέπει να έχουν ένα πολύ πιο ισχυρό στόχο στη διαχείριση αυτής της αρχής. Και μιλώ όχι μόνο για τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους, αλλά και για τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Επίσης πρέπει να δούμε τα καθήκοντα της αρχής, τα οποία θα πρέπει να συμβαδίζουν με την Ευρωπαϊκή Χάρτα το dumping θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τα πρότυπα τα οποία θα χαράξει η, Εθνική, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Δεν θα πρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας να παρεμβαίνει στο εθνικό επίπεδο. Γιατί αλλιώς θα δημιουργηθούν συγκρούσεις καθηκόντων και συμφερόντων. Επίσης, κάθε φορά που ζητάμε από τις εθνικές αρχές να αφιερώσουν χρόνο ή χρήμα για να δώσουν πληροφορίες σε μια ευρωπαϊκή αρχή, θα πρέπει να έχουμε σοβαρό λόγο, διότι φορτώνουμε τις εθνικές αρχές με έργο Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ σίγουροι για το τι ζητάμε ακριβώς και για ποιο λόγο. Δηλαδή, αυτή η διαδικασία θα πρέπει να δίνει μια προσθέμενη αξία, να βοηθάει τους πολίτες, του εργαζόμενου. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες θα δουν αυτή την προσθέμενη αξία. Αυτά ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να συζητάμε αυτό το θέμα. Thank you. Uh, Ranke from the Greens, please. Ranke, ναι, για τους πρασίνους, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εύχομαι καλή επάνωδο σε όλους μετά το καλοκαιρινές διακοπές. Προσβλέπω πάντως την θετική συνεργασία που θα έχουμε για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Όπως είπαν όλοι οι συνάδελφοι, θα πρέπει πραγματικά η αρχή αυτή να ανταποκρίνεται στο όνομα το οποίο φέρει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε αν πραγματικά η αρχή αυτή όντως μπορεί να επιβάλλει νομοθεσία, αν θα έχει την απαραίτητη εξουσία. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω σχόλια που κάναν οι προαλήσαντες, να τονίσω μόνο τρία σημεία που είναι σημαντικά για την πολιτική μου ομάδα. Κύριε Σιγητά, αναφερθήκατε στον Σέξπιρ. Θα μπορούσα και εγώ να αφερθώ στον Φάουστ λέγοντας ότι ε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ενδεχομένω και την κοινωνική ασφάλιση στο όνομα. Εμεί κάναμε την πρόταση αυτή. Είναι πολύ σημαντικό για μα η αρχή αυτή να μην ασχολείται μόνο με ζητήματα που εστιάζονται απλώ στην απασχόληση και την εργασία, γιατί αν δούμε τι κάνει το Eures, αν δούμε ποιε είναι οι διαβουλεύσει που είχε διεξάγει στο παρελθόν το Γιούρε, βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρο τη σύγχυση προκύπτει κυρίω από τα ζητήματα κοινωνική ασφάλιση και το πώ μπορούν, για παράδειγμα, στα εξωτερικά δικαιώματα να μεταφερθούν επιτυχώ από τη μία χώρα στην άλλη. Θεωρώ λοιπόν ότι μια τέτοια αρχή, σαν αυτή που θέλουμε να θεσπίσουμε, δεν θα πρέπει να ασχολείται μόνο με την κινητικό των εργαζομένων, αλλά και με τα δικαιώματα κοινωνική ασφάλιση. Όσον αφορά το ζήτημα τη ε, κατάχρηση, με κατάχρηση πολλέ φορέ έχει να κάνει με την καταχρηστική χρήση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να επικεντρωθούμε και στα προβλήματα αυτά, τα οποία πολύ συχνά αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και να μην υπάρχει μια, ένας αυθαίρετος διαχωρισμός σε διαφορετικά ζητήματα σε αυτή την αρχή. Δεύτερον, θέμα το οποίο έχουν ε, αναφέρει και διάφοροι συνάδελφοι, το ότι θα πρέπει να έχουμε όλους ενδιαφερομένους, όχι μόνο τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργοδότες, αλλά και τις οργανώσεις εκπροσώπησης της κοινωνίας των πολιτών, που πολύ συχνά γνωρίζουν ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν στην αγορά εργασίας, ιδίω διασυνοριακά σχετικά δηλαδή με την κινητικότητα διαστοριακή των εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία να συμμετέχουν και εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών. Και ένα τελευταίο σημείο, το οποίο ανέφεραν πάλι ορισμένοι συνάδελφοι, δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε εδώ πέρα έναν άνευρο, αν θέλετε, οργανισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε μέσω τη αρχή αυτή να ασκούμε πίεση, να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο διαφάνεια και να πετούμε τη διαφάνεια. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ θα πρέπει να έχουμε έναν πανευρωπαϊκό κατάλογο εταιριών, επιχειρήσεων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τον τομέα της απασχόλησης, γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε τελικά να ασκήσουμε πίεση στις επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νομοθετικές απαιτήσεις που εφίστανται σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου. δικαίου. Μόνο τότε πραγματικά μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική επιβολή της νομοθεσίας. Προσβλέπω για σε μια επικοδομητική συνεργασία μαζί σας. Δεν βλέπω εκπρόσωπο ούτε από το FTD ούτε από το ΙΕΝΕΦ, e λέει πρόεδρος. Άρα ας περάσουμε τώρα στον κατάλογο των ομιλητών. Κυρία Ρέγνερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και για μένα είναι καλή αυτή η επάνωδο. σαν να στα θρανία είναι ε, αυτή η περίοδος ε, έναρξης κοινοβουλευτική εργασίας και το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μεγάλη πρόταση ο νομοθέτης θα πρέπει να φροντίζει να ε, περνάει το δίκαιο, να ελέγχεται και να εφαρμόζεται. Αλλιώς γελιοποιείται ο νομοθέτης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και συμφωνώ με τον εισηγητή. Θα πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες, αυστηρούς και εφαρμόσιμους. Αλλά να φροντίζουμε και στη συνέχεια ότι θα λειτουργεί το σύστημα αυτό. Και ε, ε, η Ευρωπαϊκή αυτή αρχή εργασίας θα πρέπει να ε, λειτουργεί σωστά. Από την πολιτική μου δουλειά λοιπόν και την καθημερινή γνωρίζω ότι η καθημερινή διασυνοριακή συνεργασία των ε, κρατικών αρχών δεν λειτουργεί όσο ε, θα όφιλε και όπως θα θέλαμε εμείς για την εφαρμογή των κανόνων που ήδη έχουμε επιβάλει. Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών είναι πραγματικότητα και είναι και πολύτιμη αλλά εκεί παρατηρούνται διάφορα έσχη, τα είπε ο κύριος Πυρίνσκι, οι διάφορες ταχυδρομικές θηρίδες εταιρείε, ε, εικονικές, ε, θα πρέπει να καταπολεμηθούν από την ΕΛΑ. Ε, και τι χαρακτήρα πρέπει να έχει αυτή η αρχή για μένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η αρχή εργασίας να μπορεί να δρά με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγκάζει να συνεργάζονται οι εθνικές αρχές και να εφαρμόζουν τον νόμο. Αλλιώς ε, δημιουργούμε άλλη μία αρχή που θα είναι πραγματικά γελία στη λειτουργία της. Να θυμίσω λίγο και τη χρηματοπιστωτική κρίση. Τώρα έχουμε μια τραπεζική εποπτεία που λειτουργεί σωστά ε, και αντίστοιχα ε, θα πρέπει να διδαχθεί από τη συνεργασία αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Να κοιτάει πράγματα που θα είναι αρμοδιότητές της, εθνική ασφάλιση, και κοινωνική ασφάλιση και ε, να υλοποιούν σωστά όσα οφείλουν οι κρατικές αρχές. Αυτό. Thank you. Then I give the floor to Mr. Ευχαριστώ κύριο Ζορς Μπαχ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. <coughs> Πρέπει να ομολογήσω ότι σήμερα αισθάνομαι λίγο καλύτερα από ότι τον Ιούλιο. Γιατί τον Ιούλιο φαινόταν ότι ήμασταν πάρα πολύ διχασμένοι και ορισμένοι μιλούσαν και για απόρριψη. Ε, ήμασταν πραγματικά πολύ διχασμένοι. Εν περιπτώσει, εγώ είμαι πεπισμένο ότι χρειάζεται απόλυτα να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Αρχή εργασία και υποστηρίζω απολύτω τον εισηγητή μα τον συνάδελφο Γιουρούν Λέναρ. Επανειλημμένα είπαν ομιλητέ ότι αυτή η αρχή δεν θα πρέπει να είναι ωραία στα χαρτιά και μόνο, αλλά να λειτουργεί σωστά στην πράξη και να έχει τις σωστές αρμοδιότητες εξουσίας, αλλά και τα λεφτά που χρειάζεται για να λειτουργεί σωστά. Η Επιτροπή Διαμεσολάβησης δεν θα πρέπει να είναι μία επιλογή, θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί, να είναι υποχρεωτική. Επίσης πιστεύω ότι ε, χρειάζεται να συμμετέχουν περισσότερο οι κοινωνικοί εταίροι, ας πούμε στην αξιολόγηση κινδύνου, σε διάφορες αναλύσεις και να έχουμε κάθε φορά ένα εκπρόσωπο των συνδικάτων, ένα εκπρόσωπο των εργοδοτών και μάλιστα αυτή να είναι και μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ε, τέλος, θέλω να τονίσω και κάτι που είπε η Μαριάν Χάρκιν ότι εδώ δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι απέναντι στα κράτη-μέλη, αλλά να συνεργάζονται και να συμμετέχουν τα κράτη-μέλη και να υπάρχει απαραίτητη ισορροπία για να ε, έχουμε και μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για την εσωτερική αγορά και την παροχή υπηρεσιών. Το θέμα δεν είναι μόνο η ποιότητα και η ασφάλεια, αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα. Για να σταματήσει πια αυτό το κοινωνικό ντάμπινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαλάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι εισηγητής στο θέμα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνική ασφάλισης. Πολύ ακαθόδε θέμα. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας τις επόμενες εβδομάδες. Στη συζήτηση που διεξάγεται εκεί, πολύ συχνά επανέρχεται το ίδιο ακριβώ ζήτημα. το ότι δεν υφίσταται πραγματική δυνατότητα ελέγχου για την ισότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων ακριβώς επειδή δεν υπάρχει μία ε, ενιαία ευρωπαϊκή αρχή, μία ευρωπαϊκή, ένα ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς ή ένα όργανο. Η ιδέα για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ε, έρχεται να καλύψει, να συμπληρώσει ένα κενό πολύ σημαντικό και το οποίο υφίσταται σε άλλου τομεί τη κοινωνική νομοθεσίας. Η κινητικότητα των εργαζομένων ε, είναι κάτι πολύ καλό, μια πολύ καλή ιδέα, αλλά θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις απάτες, την απάτη και για να γίνει αυτό χρειάζεται μια αρχή που δεν θα είναι γραφειοκρατική. Τι είναι η γραφειοκρατία? Η γραφειοκρατία είναι όταν ε, επιβαρύνουμε τους ανθρώπους πολίτες χωρίς να εξασφαλίζουμε αποτελεσματικότητα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν καλύτερα την νομοθεσία, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τους απαταιώνες και γι' αυτό το λόγο πρέπει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία να είναι πραγματική αρχή με εξουσία. Δηλαδή οι αποφάσεις που θα λαμβάνει να έχουν αποτελεσματικότητα λένε ότι κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με τα, με την, νομοθετικά κείμενα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή Η συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. λέει το άρθρο, στο άρθρο 61 και 63 ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στο κοινωνικό τομέα. Ακριβώς γι' αυτό μιλάμε. Πρόκειται για κάτι συμπληρωματικό έναντι των εθνικών αρχών, γιατί οι εθνικές αρχές θα πρέπει να συμφωνήσουν προκειμένου να δημιουργηθεί μια τέτοιου είδους ευρωπαϊκή αρχή. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνουμε την κινητικότητα. Εγώ στηρίζω όλες τις τροπολογίες που έχουν ως στόχο να μην δημιουργηθεί μια πρόσθετη ε, αναποτελεσματική γραφειοκρατία, αλλά να είναι ένα όργανο το οποίο πραγματικά θα πρέπει να αποφάσει που θα εφαρμόζονται. Η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ. Όλοι έχουμε γυρίσει πιο δυνατοί μετά τις θερινές διακοπές. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπαλάς που λέει ότι αυτή η αρχή πρέπει να είναι αποτελεσματική, να συμπληρώνει τον, το ρόλο των κρατών μελών και των εθνικών αρχών και να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές, τους εθνικούς φορείς. Εγώ ήδη έχω υποβάλει ένα αριθμό τροπολογιών, όχι για να αλλάξουμε το όνομα της αρχής, αλλά για να διευκρινίσουμε το έργο της. Πρέπει να ξέρουμε τι χρήση θα κάνουμε αυτής της αρχής και να είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσει αντί να παρεμποδίσει. Για παράδειγμα, η χρέωση των υπηρεσιών της θα έπρεπε να αφορά μόνο τα κράτη-μέλη, όχι τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Πραγματικά πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα πρέπει να πληρώνουν για τις υπηρεσίες που θα παρέχει αυτή η αρχή δεν είναι σαφέ στην πρόταση τη Κομισιόν. Δεν νομίζω όμω ότι είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας εμεί. Επίση, εμπειρογνώμονε των κρατών μελών θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις ομάδε εμπειρογνωμόνων. Ούτε αυτό είναι σαφές από την πρόταση τη Κομισιόν. Γιατί αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, οπωσδήποτε πρέπει οι εθνικοί εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν πιο ενεργά. Οπότε χρειαζόμαστε μια αρχή που θα είναι χρήσιμη και που πραγματικά θα συντονίζει, όχι γραφειοκρατική. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, I'll give the floor to... Ευχαριστούμε. Κυρία Γιώσκοφκα, έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβλέπω όλους τους συναδέλφους εδώ πέρα, ξεκούραστους και μαυρισμένους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, με όρεξη για δουλειά. Πολλά πράγματα ήδη υπόθηκαν από τους συναδέλφους. Αναφερθώ και εγώ σε μερικά πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα θεσπιστεί αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας Ξέρετε ότι πολύ συχνά στο παρελθόν ασχοληθήκαμε με νομοθετικές προτάσεις όπου δεν υπήρχε πραγματικά ένα σκέλος ή δεδομένα όσον αφορά την απασχόληση. Ασχοληθήκαμε στο παρελθόν με την απόσπαση των εργαζομένων, με το κοινωνικό ντάμπινγκ και καταλήξαμε στο συμπέρασμα πολλές φορές ότι χρειαζόμασταν τελικά πραγματικά τον οργανισμό αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που θα θεσπιστεί αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Να δείξω λοιπόν κάποια σημεία. Πρώτον, Νομίζω ότι θα πρέπει καταρχάς να είναι σαφές πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι κοινέ επιθεωρήσεις. Οποιαδήποτε αρμοδιότητα ελέγχου θα προβλεφθεί, θα πρέπει να γίνεται από κοινού με τα κράτη-μέλη, τα εμπλεκόμενα, τα οικία κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της αναφέρεται σε μετακινούμενους εργαζόμενους. Η απόσπαση όμως των εργαζομένων έχει να κάνει προφανώς με την κινητικότητα υπηρεσιών περισσότερο παρά με την κινητικότητα της εργασίας. Ξέρουμε όμως ε, πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα των όρων απασχόληση των αποσπασμένων εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν για του όρου αυτού απασχόληση να υπάρχει μία επιθεώρηση, ένα έλεγχο και το ρόλο αυτό θα πρέπει να λάβει αυτή η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία. Στι τροπολογίε μου αναφέρομαι στο ότι η νέα αυτή αρχή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει εμπόδιο στην ευρωπαϊκή αγορά Απασχόληση. Πολύ συχνά η δική μας η Επιτροπή επιβάλλει νέα εμπόδια και φραγμούς στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αυτό ουσιαστικά αποδυναμώνει την Ευρώπη. Ξέρετε ότι ε, η δύναμη της Ευρώπης έγκυται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει ανενόχλητα να μπορούν να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης για τους ε, Ευρωπαίους εργαζόμενους. Απευθύνουμε λέει, τώρα πρόεδρο στην... στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ετέθησαν κάποια ερωτήματα, ενδεχομένω να θέλετε κι εσείς να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την εργασία που έχετε επιτελέσει μέχρι σήμερα. Ξέρω πόση δουλειά κρύβεται πίσω από τις τροπολογίες αυτές, πόσες συνεδριάσεις χρειαστήκατε να κάνετε. Ξέρουμε ότι ανέκαθεν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξο όσον αφορά την πρόταση αυτή και βλέπουμε ότι πραγματικά ανταποκρίνεται στην αρχική του αυτή φιλοδοξία. Επί του παρόντος δεν μπορούμε εμείς να σχολιάσουμε τις τροπολογίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν εγκριθεί. Ενδεχομένως θα μπορούσα να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα και να επαναλάβω κάποια σημαντικά στοιχεία της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως και περισσότερο, έτσι και εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε έναν λειτουργικό οργανισμό, μια καλώς λειτουργούσα αρχή, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει προφανώς να δίδει περισσότερες πληροφορίες, να μεσολαβεί, να συνεργάζεται και να συντονίζει τη δράση των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να παρέχει πληροφορίες, να ενισχύει τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές και θα πρέπει επίσης η αρχή αυτή να έχει τη δυνατότητα να προβλέπει και κάποιες λύσεις μέσω της διαμεσολάβησης. Αυτό ακριβώς προτείνουμε, σε αυτό ανταποκρίνει τη δέσμη μέτρων που έχουμε υποβάλει Προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε μία αρχή η οποία να μπορεί να συμπεριλαμβάνει όλες αυτές τις διαφορετικές λειτουργίες. Όσον αφορά τώρα το όνομα της αρχής αυτής, ξέρετε ότι και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάναμε πολλές συζητήσεις. Προφανώς η αρχή αυτή θα ασχοληθεί με την ελεύθερη κινητικότητα των εργαζομένων, με την κοινωνική ασφάλιση, με την απόσπαση των εργαζομένων. Θεωρούμε ότι όλες αυτές οι διαστάσεις ε, αποκρισταλώνονται σωστά στην ε, προτινόμενη ονομασία Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία και έτσι προκύπτει στα αγγλικά και το αρχικό ELA, ένα αρχικό το οποίο δεν χρησιμοποιούσαμε. Βλέπω ότι ε, ένα βασικό ρόλο που προβλέπεται για την αρχή αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παροχή πληροφοριών, δηλαδή αφισβητείται αυτή τη στιγμή από κάποιου ευρωβουλευτέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω να διατηρήσουμε το ρόλο αυτό αυτή τη αρχή, την παροχή δηλαδή πληροφοριών, γιατί αυτό θα καταστήσει τελικά την αγορά εργασία πιο συνεκτική, θα βοηθήσει τόσο του εργοδότε όσο και του εργαζόμενου και θα προωθήσει ακόμα περισσότερο την κινητικότητα των εργαζομένων. Ένα από εσά αναφέρθηκε σε μια ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Προφανώ την έκθεση αυτή την έχουμε λάβει πολύ σοβαρά υπόψη μα. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στι συστάσει του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και θεωρούμε ότι θα πρέπει να σταματήσει πλέον ο κατακρεματισμό που είχαμε δει στο παρελθόν όσον αφορά την παροχή πληροφοριών για την αγορά εργασία και να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία θηρίδα, έναν οργανισμό ο οποίο θα μπορεί να παρέχει αυτέ τις πληροφορίες παράλληλα με τις ε, υπόλοιπες, ε, τα υπόλοιπα καθήκοντα τα οποία θα επιτελεί. Είμαστε σε επαφή με του κοινωνικού εταίρου, το επαυτό ένα άλλο Ευρωβουλευτή, δεν του ξεχάσαμε, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο ζήτημα τη κινητικότητα των εργαζομένων, τη ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και γι' αυτό ακριβώ το λόγο προβλέπουμε στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα υπάρχει αυτή η ομάδα ενδιαφερομένων στα πλαίσια τη οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών. Ολοκληρώνω την παρέμβασή μου στο σημείο αυτό, και είμαι προφανώ στη διάθεσή σα για επιπλέον ερωτήσει ή άλλε παρατηρήσει που ενδεχομένω ε, να έχετε. Είμαι στη διάθεση τη δική σα και όλο ιδιαίτερο βέβαια στη διάθεση του εισηγητή και τη ομάδα του. Σα ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά για όλη την εργασία την οποία έχετε επιτελέσει και το γεγονό ότι καταφέρατε πραγματικά να τηρήσετε αυτό το τόσο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα το οποίο είχατε προτείνει στην αρχή τη όλη διαδικασία, Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε τότε το λόγο στον ε, εισηγητή μας, τον κύριο Λένερς, ο οποίος ενδεχομένως να έχει και κάποιες ερωτήσεις εξ ονόματος Επιτροπής μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε και αυτές να τις θέσετε. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω να θέσω ερωτήσεις αυτή τη στιγμή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλου του αδέλφου για την αφοσίωσή του, για τη δέσμευσή του. Όπω είπε και ο κύριο Μπάχα, σιγά σιγά κινούμεθα προ ένα κοινό σημείο σύμβλεψη όσον αφορά την πρόταση αυτή. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να διευθετήσουμε λίγο περαιτέρω όσον αφορά την παροχή πληροφοριών. Δεν θα ήθελα να υπάρχει επ' αυτού κάποια παρεξήγηση. Και εγώ πιστεύω ότι η παροχή πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ προέρχομαι από μία μεθόρια περιοχή στα σύνορα πολύ κοντά με μια άλλη χώρα, συνειδητοποιώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν πληροφορίε όσον αφορά την διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων. Οι πληροφορίε αυτέ δεν θα πρέπει αναγκαστικά όμω να παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έλαβα μάλιστα πολλά emails και επιστολέ από τους ψηφοφόρους μου σε εβδομαδιαία βάση, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το φορολογικό συντονισμό. Καταλαβαίνετε ότι επί των ζητημάτων αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Πώς θα καταφέρει ποτέ η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας να παρέχει τόσο λεπτομερείς λεπτο, ε, πληροφορίες εθνικής φύσης τελικά όσον αφορά την ε, εργασιακή νομοθεσία, όσον αφορά την ε, κινητικότητα των εργαζομένων και πώς θα καταφέρει ουσιαστικά να τους δώσει πληροφορίες που είναι καθαρά διμερείς. Για παράδειγμα, συμφωνίες φορολογικές που μπορεί να έχει συνάψει η Γερμανία με κάποιες άλλες όμορες της χώρες. Νομίζω ότι οι πληροφορίε αυτέ σαφώ θα πρέπει να παρέχονται στου εργαζόμενου, αλλά δεν θα πρέπει να δίδονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ζήτημα αυτό μπορεί να διευθετηθεί πολύ αποτελεσματικά σε διμερέ εθνικό επίπεδο. Για όλα τα υπόλοιπα σχόλια βλέπω ήδη ότι έχει περάσει η ώρα. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε ασχοληθεί αρκετά με το ζήτημα αυτό. Προσβλέπω σε μια θετική συνεργασία με όλους τους συναδέλφους κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώ ευχαριστώ πολύ και εγώ για όλες τις παρεμβάσεις σας. Χρονοδιάγραμμα. Εμείς εδώ θα ψηφίσουμε στις 18 Οκτωβρίου στην Ολομέλεια. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα πάει, δεν έχει αποφασιστεί. Προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Ορίστε. Δεν έχουμε τον εισηγητή. Κανονικά θα πρέπει να προχωρήσουμε στο σημείο 8, αλλά αποσιάζει ο εισηγητής ο κύριος Καλβέτ Σαμπό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του και η έκθεση που θα συζητήσουμε. Να περιμένουμε πέντε λεπτά. Δεν ξέρω αν θέλει να ξαναμιλήσει κανείς για κάτι άλλο. Για την αρχή εργασίας. Δέκα, πέντε λεπτά. Μη φύγετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα 8 για το Κοινοβούλιο.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 pour... C'est ça, c'est au long terme. Parce qu'évidemment, il faut... Oui, c'est convaincre. OK, friends, uh, let's... Ωραία, λοιπόν. Φίλοι, ας ξαναρχίσουμε. Συνεχίζουμε το σημείο 8 στη μέση διάταξη διαφανής και προβλέψιμη όρη εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. And, uh, I'll start Θα δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Καλβέ Σαμπόν και μετά θα ακολουθήσουν οι σκιώδεις εισηγητές και τα λοιπά μέλη που θα έχουν σίγουρα να κάνουν σχόλια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Παρακαλώ. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλή επιστροφή. Καλώς όρισαν όλοι όσοι επέστρεψαν από αυτές τις μακρόχρονες τερινές διακοπές. <clears throat> Θα μιλήσω στα ισπανικά, εκτός και αν απαντήσω κάποιες ερωτήσεις. Πρόκειται για μια οδηγία πολύ ευαίσθητη και χρειάζεται να είμαι ακριβής, γι' αυτό το λόγο έχουμε και τους διερμηνείς. Το πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα σε αυτή την οδηγία μας πιέζει. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Διότι η Κομισιόν αλλά και όλοι ε, επιθυμούν αυτή η οδηγία να υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας. Πριν δηλαδή ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία. γιατί μπορεί να έχει πολύ θετικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την εικόνα του Κοινοβουλίου στην κοινωνία. Η κοινή γνώμη δίνει ιδιαίτερη σημασία σε, αυτή την, αυτό το θέμα. Ε, πρόκειται για μία από τις πρώτα, από τα πρώτα, ένα από τα πρώτα νομοθετικά κείμενα που προκύπτουν από τον κοινωνικό πυλώνα μετά την ε, συμφωνία του Γκέτεμπορκ. Βλέπω ότι και οι συνάδελφοί μου με τους οποίους συνεργάζομαι κατανοούν αυτή τη σημασία και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Έχοντας διαβάσει όλες αυτές τις τροπολογίες, μεγάλο αριθμό, ε, τροπολογιών οι οποίες δείχνουν ότι το θέμα ενδιαφέρει τους συναδέλφους. Μπορώ να πω το εξή. Τα κεφάλαια τα οποία πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε σημεία ισορροπίας και που δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα απόλυψης οδηγίας είναι το ε, κεφάλαιο πληροφόρησης για τις ερασιακές σχέσεις Εκεί υπάρχει δυνατότητα να συζητήσουμε το πότε θα δίδονται οι πληροφορίες, πότε θα δίδεται η πληροφόρηση σε σχέση με την ευαισθησία που πρέπει να δείξουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το διοικητικό άχθος. Με ευελιξία, στις συναντήσεις μου έμαθα ότι η πληροφορία της πρώτης ημέρας είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, κάτι που δεν το ήξερα. Μπορούμε λοιπόν να ε, προσαρμοστούμε έξυπνα στην πραγματικότητα ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των, μικρο, μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές ή που δεν χειρίζονται καλά το ίντερνετ θα πρέπει να δώσουμε μια ευελιξία. Δεν νομίζω ότι εκεί θα αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα. Για τα δικαιώματα, επίσης. Μια, ο μια μιας σε μία ενδιάμεση ημερομηνία σε ό,τι αφορά την δοκιμαστική περίοδο. Είναι κάτι εφικτό. Βέβαια, το καλύτερο είναι εκτός του καλού. Οπότε πρέπει η οδηγία αυτή να δίνει συγκεκριμένα μηνύματα και τα αποτελέσματα. Γιατί απευθυνόμαστε στους πολίτες μας και πρέπει να τους πούμε, για παράδειγμα, αν πούμε ότι η μέγιστη, περίοδος, η μέγιστη διάρκεια τη δοκιματική περίοδου είναι το 25% της, ε, του χρόνου τη σύμβαση. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο για τους πολίτες. Νομίζω ότι και εκεί θα βρούμε κάποια ισορροπία με ε, αμοιβές παραχωρήσεις. σίγουρα δεν θα είμαι μαξιμαλιστής. Μετά υπάρχει το θέμα της τροποποίησης, βελτίωσης της εργασιακής σχέσης που θα δημιουργήσει ένα δικαίωμα και θα πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένα κανάλια για να γίνεται κάτι τέτοιο. Μετά, πληροφόρηση των αποσπασμένων εργαζομένων. επιπλέον των όσων ήδη προβλέπονται. Δεν έχω πρόβλημα με αυτά. Εκεί νομίζω θα βρούμε λύση. Ισορροπημένη λύση. Δεδομένου ότι η εργασία που έχει κάνει η Κομισιόν είναι πολύ καλή. Οι ελάχιστες απαιτήσει. Παρόμοιο ζήτημα. Ο, παρόμοιο με αυτό των δικαιωμάτων. θέματα που μπορεί να συζητήσουμε. Ποια είναι. Οι εργοδότες ζητούν να μην είμαστε υπερβολικά αυστηροί διότι θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Θα πρέπει αυτό να το εξορροπήσουμε με το να μην δημιουργήσουμε κερκόπορτες, παραθυράκια που θα οδηγήσουν, θα επιδώσουν το, τη δυνατότητα στους εργοδότες να παρακάμπτουν χωρίς έλεγχο και επαορίστο τους κανόνες. Για παράδειγμα, συμβάσεις μηδενικής διάρκειας. Πάντοτε έλεγα ότι δεν θα λύσουμε εδώ το ζήτημα του κατά πόσον αυτές οι συμβάσεις θα πρέπει να απαγορεύονται ή όχι. Όχι, δεν είναι αυτή η πρόθεση. Όμως μπορούμε να πάρουμε μέτρα κοινή λογικής με βάση τα όσα εμείς στην Ευρώπη θεωρούμε εργασιακή ή συμβατική σχέση. Έτσι ώστε αυτό, αυτή η έννοια να μην επιτρέπει μ, ε, παρεκτροπές μέσω των συμβάσεων μηδενικής διάρκεια. Τούτου λεχθέντο. Αυτό που πραγματικά είναι προβληματικό και διχάζει πραγματικά τις τροπολογίες που έχω λάβει είναι το θέμα των ορισμών, το θέμα του τι είναι εργαζόμενος. Ε, μια νοσοκόμα και το ε, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν δύο πράγματα για αυτό και εκεί έχουμε κολλήσει. Εκεί αυτό είναι το προβληματικό ζήτημα. Πρόθεση του κειμένου είναι να αναγνωρίσει ότι οι πολίτες έχουν μια σειρά δικαιωμάτων όταν εργάζονται, όταν βρίσκονται στον, ε, στον κόσμο της εργασίας, που χαρακτηρίζουν τον Ευρωπαίο εργαζόμενο και που θα πρέπει να τα μπορεί να, μπορεί να τα ασκήσει ανεξαρτήτως της νομικής μορφής εργασιακής σχέσης που τον διέπει. Εγώ αυτό που βλέπω είναι μια διπλή ανησυχία. Αφενός, κάτι το οποίο συμμεριζόμαι απόλυτα, κανείς δεν πρέπει να μείνει εκτός αυτών των δικαιωμάτων. Πρόκειται για καθολικά και ευρωπαϊκά δικαιώματα. Κανείς εργαζόμενος ή και κανείς από αυτούς που έχουν εργαστεί στο παρελθόν δεν πρέπει να στερηθεί τα δικαιώματα αυτά. Αυτό αφενός. Αφετέρου τώρα υπάρχει μια άλλη ανησυχία πιο τεχνική και νομική, έχει σχέση με ε, την εκπαίδευση που έχουν λάβει οι, αυτοί που έχουν υποβάλει τις, εργοδο... Ε, τροπολογίες. Ε, δεν θα πρέπει, λένε, να επηρεαστούν τα συστήματα δικαίου των κρατών μελών, αρχή της επικορικότητας κλπ. κλπ. Θα πρέπει, πιστεύω εγώ προσωπικά, να ξεφύγουμε από αυτό το σκόπελο θα πρέπει να εστιάσουμε στα δικαιώματα και όχι στην νομική εφαρμογή και στους νομικούς κώδικες. Εγώ θα κάνω μια γραπτή πρόταση όπου θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στην ουσία. Ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι κάθε άτομο, δεν μιλώ για εργαζόμενο μόνο, κάθε πολίτης που εξαρτάται οικονομικά, εξαρτάται οργανωτικά, εξαρτάται λειτουργικά, ιεραρχικά. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, κάθε τέτοιο άτομο, κάθε τέτοιος πολίτης να καλύπτεται από αυτά τα δικαιώματα. Και μετά, κάθε χώρα αναγκαστικά κάθε χώρα θα εφαρμόσει αυτά τα δικαιώματα σύμφωνα με τη δική της εργασιακή νομοθεσία. Και λέω κάθε χώρα διότι δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Και τι εννοώ με αυτό. Κάθε χώρα μπορεί να μιλάει για εργαζόμενους, ε, ελεύθερους επαγγελματίες, ψευδοελεύθερους επαγγελματίες κλπ. κλπ. Δεν έχει σημασία πώς, τι ορισμό δίνει. Αυτός όμως ο οποίος εξαρτάται οργανωτικά, διοικητικά, ιεραρχικά κλπ. από κάποιον εργοδότη καλύπτεται. Όπως και να τους ονομάζουμε. κάθε χώρα θα δώσει το δικό της ορισμό. Θα πρέπει όμως αυτά τα δικαιώματα να καλύπτουν όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η πρότασή μου, διότι αν αρχίσουμε και μιλάμε για τον πραγματικό ορισμό του εργοδότη, του εργαζόμενου από νομικής πλευράς, θα αρχίσουμε να ακούμε αντιρρήσεις και διαφωνίες διότι κάποιοι θα αισθανθούν ότι πλήττονται τα παραδοσιακά του ε, συστήματα κλπ. Εγώ αυτό που θέλω είναι απλώ κάθε χώρα θα πρέπει να προσαρμοστεί τελικά σε μια οδηγία δικαιωμάτων. Όχι βασική οδηγία, οδηγία δικαιωμάτων. Θα πρέπει τελικά τα δικαιώματα αυτά να προσαρμοστούν στις νέες μορφές εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοδοξία της Ευρώπης. Αυτά μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να ξεσκονίσουμε την άμμο από πάνω μας και να σηκώσουμε τα μανίκια. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο εκπρόσωπός του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ εισηγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θέλω να πω ότι έχω εκνευριστεί λίγο και για να μην πω ότι ε, έχω θυμώσει. Κανονικά προβλεπόταν το θέμα αυτό για το απόγευμα και το είχα γράψει και στην ατζέντα μου. Και ξαφνικά το βάζετε και μετά το καλοκαίρι ε, άρων-άρων το πρωί και χρειάστηκε να φύγω από ένα άλλο ραντεβού και μια υποχρέωση που είχα. Πραγματικά αυτό δεν ανταποκρίνεται ούτε στη σημασία ούτε στο αντικείμενο το ίδιο και στο ύψος των περιστάσεων και θα ήθελα να το πω. Ε, κατά τα άλλα, Συμφωνώ λίγο και με την αισιοδοξία του εισηγητού. Το ε, είδαμε αυτό και κυριάρχησε μέχρι τώρα συζητήσεις των σκιωδών εισηγητών. Υπάρχει ευρύτατη συναντήληψη ε, και ομοφωνία για το θέμα αυτό το θέμα δεν είναι να κάνουμε έτσι ένα λυρικό κείμενο με κοινωνική πολιτική για φιλολογία, αλλά ε, να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σε μερικά σημεία πραγματικά πιστεύω ε, ότι είμαστε σε καλό δρόμο, ωστόσο πρέπει να πω και με κάθε σαφήνεια και να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχουν και μερικά σημεία ε, όπου απέχουμε έτη φωτός από το συμβιβασμό και δεν βλέπω να συμβιβαζόμαστε και να τα βρίσκουμε. Ε, παράδειγμα τώρα, ε, η νομικός ορισμός του εργαζομένου. Εμένα μου αρέσει πολύ η άποψη του εισηγητού και βλέπω με συμβάθεια που λέει ας σταματήσουμε τα νομικίστικα και να ασχοληθούμε με την ουσία της πολιτικής. Ωραία είναι αυτά, αλλά... Ε, ε, για κάποιον που δεν είναι νομικό, καλό είναι να μην αναλόμαστε στα δικηγορίστικα γιατί λιγότερα νομικά σημαίνει περισσότερη κοινή λογική αλλά επειδή είμαστε και κοινοβούλιο τα νομικά έχουν σημασία ιδιαίτερα για τη μεταφορά του δικαίου στα κράτη-μέλη γιατί ε, δεν μπορούμε σε ένα τέτοιο θέμα να εξαιρέσουμε τελείω τη νομική διάσταση ε, Πού το πάω. Να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στα θέματα που συμφωνούμε για να ξεκαθαρίσουμε και πριν τις εκλογές ότι τα δικαιώματα και τα, τα θέματα των εργαζομένων δεν μας είναι καθόλου αδιάφορα. Ενώ σε θέματα που δεν διαφαίνεται συμβιβασμό, όπως αυτό που σας είπα τώρα, το νομικό ορισμό της έννοιας ε, του εργαζομένου, θα πάμε να συγκρουστούμε στην ψηφοφορία και με μια ε, πλειοψηφία θα περάσει η α ή β άποψη. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό τώρα για να ε, παραγωνιστούν τα μεγάλα και τα πολλά που μας ενώνουν. Συνεχίζεται λοιπόν αυτή η συζήτηση για να δούμε πάντα πώς θα προωθήσουμε τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόπεθ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία όλων αυτών των μηνών που κάναμε για να φτάσουμε ως εδώ και ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές όλοι μαζί. Συμφωνώ με ε, όσα υπόθηκαν ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες να προχωρήσει και να προωθήσει μια νομοθεσία εργασιακή γιατί είναι πολύ σημαντική. Αυτό σημαίνει τη μεταφορά στην πράξη και σε νόμο αυτή τη θαυμάσια ιδέα που είχε και το Κοινοβούλιο για τον κοινωνικό πυλώνα, αλλά τώρα θα πρέπει επιτέλου να προσγειωθεί στην νομοθεσία. Ε, έχουμε ε, τις αλλαγές ε, στην κοινωνία μας, στην εργασία μας, τα οικονομικά προβλήματα και θέματα αναδιανομής του πλούτου. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αγορά εργασίας και τις αλλαγές που γνωρίζει. Γι' αυτό έχουμε και μια τέτοια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έρχεται τούτων λεχθέντων πρέπει να πω ότι είναι αγαστή η συνεργασία και ευχάριστη όλων των πολιτικών ομάδων και χάρη στον εισηγητή. Τέσσερις είναι μεγάλοι τομεί διαπραγμάτευσης. Δύο θέματα μεγάλα που έχουν να κάνουν με τα ελάχιστα κατώτερα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στι εργασιακέ συνθήκες και οι δέσμοι των πληροφοριών Εκεί βρίσκουμε χώρους συνεννόηση με φυσικό τρόπο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει καλή πρόταση. Και μετά από τις διάφορες θέσεις που υπάρχουν κάπου θα ε, τα βρούμε. Από την άλλη μετά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο επίσης σημαντικό για τη δική μας πολιτική ομάδα και αυτό είναι το άρθρο 12 της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την αναγνώριση και την προστασία ορισμένων εργασιακών ε, μοντέλων σε κάποια κράτη-μέλη που βασίζονται στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις και αυτά λειτουργούν σωστά. Και προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτεθεί αυτή την οδηγία, αλλά θα πρέπει να τα αναγνωρίζει αυτά τα δικαιώματα και να τα προστατεύει, ιδιαίτερα στις βορειοευρωπαϊκές χώρες. Και θα πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτό ότι ε, ε, μιλάμε για ελάχιστες εργασιακές συνθήκες και προδιαγραφές, αλλά θα πρέπει να προστατεύουμε και αυτά τα μοντέλα. Και αυτό είναι δική μας δέσμευση, πολύ σημαντική, των σοσιαλιστών και δημοκρατών, αλλά και των άλλων πολιτικών ομάδων, για να δούμε πώς θα ε, μεταφραστεί σε συγκεκριμένο κείμενο. Και το τέταρτο και τελευταίο στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όπως πολύ σωστά είπε και ο εισηγητής, αλλά και προηγουμένως ακούσαμε ότι δίστανται απόψεις και σημαντικά, είναι ε, ορισμό στο άρθρο 2. Εμείς σοσιαλιστές και δημοκράτες τι θέλουμε να πούμε ως ομάδα. Αυτό που έχει για μας σημασία και στη διαπραγμάτευση δεν είναι να είμαστε τίποτα ιερείς της ευρωπαϊκής κωδικοποίησης για τα εργασιακά δικαιώματα, για να κωδικοποιηθεί τι είναι το ευρωπαϊκό ε, δικαίωμα ή και ο Ευρωπαίος Για μας έχουν σημασία τρία πράγματα στην οδηγία. Πρώτον, το πεδίο εφαρμογή. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερον, η ασφάλεια δικαίου, οπωσδήποτε, ε, την οποία θα πρέπει να επιφέρει. Και το τρίτο είναι η επιβολή της οδηγίας. Enforcement το λένε αυτό στα αγγλικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και όχι μόνο για τον ορισμό αλλά και για τα συμφέροντα που υπάρχουν από πίσω και τα τρία αυτά στοιχεία γιατί από εκεί θα εξαρτηθεί εάν θα καταφέρουμε η οδηγία αυτή να καλύπτει πολύ κόσμο, να καλύπτει νέα φαινόμενα στην αγορά εργασίας όπως είναι οι ψεύδο αυτοαπασχολούμενοι με τις νέες πλατφόρμες και νέες μορφές στην αγορά εργασίας που παραβιάζουν αυτή την ε, συγκεχημένη διαχωριστική γραμμή για το πότε είσαι εργαζόμενος και πότε εργοδότης, επιχειρηματίας δηλαδή, στην πράξη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς. Να προχωρήσει η οδηγία με καλό συμβιβασμό, να δεσμευτούμε ότι θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και ότι η οδηγία θα προστατεύει και θα σέβεται διάφορα εργασιακά μοντέλα στην Ευρώπη, αλλά θα βάνει υπόψη και τις αλλαγές, τις επισφαλείς μορφές εργασίας, τις νέες μορφές εργασίας που είναι πιο ασαφείς και πιο συγκεχημένες, αλλά που και εκεί χρειάζεται προστασία από τη συγκεκριμένη οδηγία. Thank you. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Μακιντάρη, εξ του ECR. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Τον ευχαριστώ ειλικρινά για όλη αυτή την προσπάθεια που έχει καταβάλει στη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Πραγματικά εκτιμήσα πάρα πολύ την αγαστή συνεργασία που είχαμε και το ότι έλαβε υπόψη του όλες τις ανησυχίες μας, καθώς επίσης και όλα τα σημεία εκείνα που εμείς θεωρούσαμε σημαντικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή για τον τρόπο εργασίας, που είχαμε και θεωρώ ότι πραγματικά θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική συμφωνία. Υπάρχουν διάφορα σημεία από των οποίων θα ήθελα να κάνω τώρα κάποια σχόλια. Πρώτον, μου προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, θα έλεγα, η πρόταση του Συμβουλίου να αποκλείσει τις δημόσιες υπηρεσίες και όσους εργάζονται στις δημόσιες υπηρεσίες από την οδηγία αυτή. Πραγματικά δεν υπάρχει καμία δικαιολόγηση για κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ενδεχομένως ε, κάποιες υπηρεσίες όπως οι ένοπλες δυνάμεις να έχουν διαφορετικές απαιτήσει. Ενδεχομένως. Αλλά από την άλλη μου φαίνεται περίεργο το Συμβούλιο να θέλει να αποκλείσει πραγματικά όλους όσοι εργάζονται σε κυβερνητικού οργανισμού στο δημόσιο τομέα. Είναι συναλλή ουσιαστικά το Συμβούλιο ότι δεν υποστηρίζει την ίδια την οδηγία. Αν λοιπόν έρχονται τα ίδια τα κράτη-μέλη και λένε πολύ ωραία, αυτά ισχύουν για όλου του άλλου, αλλά όχι του δικού μα του εργαζόμενου, αυτό στέλνει ένα πολύ λαθασμένο μήνυμα. Θεωρώ ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να πει ξεκάθαρα ότι η οδηγία αυτή θα εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο και στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Επομένως θα πρέπει να λάβει πιο σοβαρά την πρόταση αυτή το ίδιο το Συμβούλιο και να πει ξεκάθαρα και ρητά ότι θα εφαρμόζεται τόσο στους υπαλλήλους του ιδιωτικού όσο και στους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Πρώτη παρατήρηση αυτή. Δεύτερον τώρα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλος στόχος αυτής της πρότασης οδηγίας είναι να δημιουργήσει ελάχιστα δικαιώματα προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια και προβλεψιμότητα στις εργασιακές σχέσεις. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερε προσπάθειε, να βελτιώσουν την κατάσταση, την εργασιακή και αυτό συνάδει απόλυτα με τη δική μα τη γραμμή. Πάντα ξέρετε ότι οι οδηγίε δημιουργούν ελάχιστα πρότυπα και έρχονται τα κράτη-μέλη εν συνεχεία και προσαρμόζουν την οδηγία αυτή, ενδεχομένω τη βελτιώνουν κάθε φορά την προσαρμόζουν στις εθνικές περιστάσεις. Αυτό σημαίνει για μα ότι δεν πρέπει να προβλέψουμε τα πάντα εκ των προτέρων, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια πάρα πολύ καλή βάση. Το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο προκύπτει για μένα είναι η χρήση του όρου εργαζόμενους. Ενώ νομίζω ότι ουσιαστικά θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο απασχολούμενος, μισθωτός. Ξέρετε ότι έχουμε εργαζόμενους σε διάφορες μορφές εργασίας, όπως σε πλατφόρμες για παράδειγμα, αλλά αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή στην οδηγία αυτή είναι να, να καθορίσουμε τη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι μισθωτοί. Επομένως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι και από την άλλη πλευρά, για παράδειγμα για τους εργοδότες, δεν αναφερόμαστε σε αφεντικά σε προσταμένου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν από την μία πλευρά να έχουμε σαφή αναφορά στους εργοδότες, σαφώς, και από την άλλη πλευρά να χρησιμοποιείται τουλάχιστον στα αγγλικά όρος employee και όχι worker, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί θεωρώ ότι κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε έναν ορισμό πολύ πιο συγκεκριμένο. Καταλαβαίνω ότι ε, θα πρέπει να καλύψουμε εργαζόμενους με διαφορετικές ε, μορφές εργασίας. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την επέκταση του ε, ορισμού employee στα αγγλικά. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο όρος worker, ο οποίος είναι αρκετά ασαφής και δεν είναι νομικά δεσμευτικός. Ξέρουμε ότι οι εθνικοί ορισμοί έχουν προσαρμοστεί τα τελευταία χρόνια το εργατικό δίκαιο, οι συλλογικέ συμβάσει, η σχετική εθνική νομολογία έχει λάβει υπόψη τι όλε τι αλλαγέ που έχουν γίνει στο εργατικό δίκαιο και στην, στα συστήματα κοινωνική ασφάλεια. Τώρα, ένα άλλο τομέα που απασχολεί είναι ότι η οδηγία αυτή προσπαθεί να μην καλύψει τομεί που έχουν καλυφθεί από άλλε οδηγίε. Αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να είναι ο στόχο μα. Έχουμε, για παράδειγμα, μια, υπηρεσία, έχουμε μια οδηγία όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων. Έχουμε μια άλλη οδηγία όσον αφορά του προσωρινά απασχολούμενου. Α μην προσπαθήσουμε μέσω τη οδηγία αυτή να καλύψουμε τομεί του οποίου ήδη του έχουμε καλύψει, ήδη του έχουμε διευθετήσει με άλλα νομοθετήματα. Και το λέω αυτό γιατί ω εργοδότης. Όταν ε, προσπαθεί κανείς να συμμορφωθεί με την νομοθεσία αυτή, πολλές φορές βρίσκεται αντιμέτωπο με κάποια αντιφατικά σημεία. Υπάρχει, για παράδειγμα, μια οδηγία για την απόσπαση του εργαζομένου, για παράδειγμα, που μπορεί να προβλέπει συγκεκριμένε διατάξεις. Και έπειτα προσκρούει κανείς σε μια άλλη ευρωπαϊκή οδηγία, ενδεχομένω να λέει κάτι το αντιφατικό είναι πάρα πολύ σημαντικό στον τομέα του εργατικού δικαίου οποιαδήποτε οδηγία εμείς εγκρίνουμε να μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από το μικρό επιχειρηματία ο οποίος προσπαθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να γίνει ένας καλός εργοδότης. Α μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίε οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή την πληθώρα των διαφορετικών νομοθεσιών που έχουμε εγκρίνει. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί εύκολα και γρήγορα ένα δυνητικό επιχειρηματία να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να είναι καλό εργοδότη. Και έχω καταθέσει και μία επιπλέον τροπολογία όσον αφορά τι διατάξει εκείνε που έχουν να κάνουν με την κατάρτιση. Γι' αυτό διότι θα ήθελα να αποτρέψουμε αυτή την πρακτική που στα αγγλικά ονομάζεται pay to fly, το οποίο είναι πρακτική που έχει να κάνει για παράδειγμα με πιλότες οι οποίοι αναγκάζονται οι ίδιοι να πληρώσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης προτού απασχοληθούν σε μια επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή προφανώς θα πρέπει ο εργοδότης να χρηματοδοτεί την κατάρτιση εν προκειμένου του συγκεκριμένου πιλότου σε ένα αεροσκάφος. Ήθελε λοιπόν και το σημείο αυτό να συμπεριληφθεί προκειμένου να μην έχουμε τέτοιες ε, πρακτικές και τουλάχιστον σας ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε για τον φάκελο αυτόν. Σας ευχαριστούμε. Τώρα η κυρία Παλώμα Λόπεθ Μπερμέγιο έχει το λόγο εξ ονόματο της ΓΚΟΕ. Παρακαλώ. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του και για τις ειλικρινείς προσπάθειες που καταβάλει να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο. Επίσης να ευχαριστήσω τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές. Οι διαπραγματεύσει ξεκίνησαν πριν το καλοκαίρι, είναι νωρί ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά να υπογραμμίσω ότι βλέπουμε μια σαφή διάθεση συμβιβασμού από όλου. Και αυτό είναι πολύ καλό. Με τον εισηγητή συμμερίζομαι την ανάγκη η όλη διαδικασία να επιταχυνθεί έτσι ώστε να, ολοκληρω, να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ε, τρέχουσας θητείας. Θέλω να υπογραμμίσω ορισμένα ζητήματα σε σχέση με τα όσα έχουμε πει ως τώρα και όσα έχω ακούσει. Κάποια άλλα βέβαια στοιχεία θα τα αφήσω για αργότερα, για τις επόμενες συναντήσεις μας. Όπως έλεγα λοιπόν, για μας είναι πολύ σημαντικό κανείς εργαζόμενος να μην εξαιρεθεί από τα δικαιώματα της οδηγίας. Θα δούμε σε λεπτομέρειε το πεδίο εφαρμογή, αλλά ήδη προκύπτουν ορισμένα ζητήματα σε σχέση με τον αποκλεισμό εργαζομένων. Σημείο κλειδί είναι η δοκιμαστική περίοδος. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να το λύσουμε, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του χρόνου εργασία του κλπ, θα πρέπει να έχουν δικαίωμα τα ίδια δικαιώματα μάλλον που αναφέρονται, που αναφέρονται στην οδηγία μεταξύ αυτών και την προστασία που, καλύπτεται, που τους καλύπτει. Η διάρκεια της δοκιμαστικής περίοδου θα πρέπει να είναι ανάλογη της εργασιακή σχέσης και του επαγγέλματο, αλλά δεν είναι δυνατόν να έχει μια διάρκεια υπερβολική. Προτείνουμε ποτέ να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες στα πιο απαιτητικά επαγγέλματα. Πάντως θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η διάρκεια της και όλοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα και την ίδια προστασία. Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση, την επιμόρφωση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται μέσα στο ωράριο εργασίας και θα επιμείνουμε σε αυτό. Όλη η επιμόρφωση που είναι υποχρεωτική για τον εργαδότη και τον εργαζόμενο. Και βέβαια προφανώ να μην χρειάζεται να πληρώνει ο εργαζόμενο για να ε, λάβει αυτή την επιμόρφωση. Άλλο σημείο. Η ρήτρα μη επιστροφής. Πέραν των όσων ήδη αναφέρονται, θέλουμε να υπογραμμίσουμε και να επιμείνουμε ότι κανείς εργαζόμενος δεν θα δει τις συνθήκες εργασίας του να χειροτερεύουν μετά την ε, υιοθέτηση της οδηγίας. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί αυτή η ρήτρα της ε, μη επιδείνωσης, να το πούμε έτσι καλύτερα. Μετά μας ε, ανισχύει το θέμα των ορισμών. Πράγματι, έχουμε καινούριες μορφές εργασίας, με πολλά καινούρια στοιχεία, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Αν πετύχουμε με τον ορισμό, τότε οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες ε, δεν θα μείνουν εκτός του ορισμού και συνεπώς δεν θα μείνουν προστάτευτοι. Εμένα αυτό που πιο πολύ όμως με απασχολεί είναι ο ορισμός του εργοδότη, όχι του εργαζόμενου. Γιατί είναι πολύ σημαντικός ο ορισμός αυτός για τον καθορισμό των σχέσεων το πόσο είναι ένας ή πλίονες οι εργοδότες σε κάθε περίπτωση. Και αν δεν το καταφέρουμε, δεν να δώσουμε το σωστό ορισμό, μπορεί να δημιουργήσουμε νομικά κενά και ασάφειες. Τελειώνω λέγοντας ότι για μας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες ε, σε αληφτικά σκάφη και ως οικιακό προσωπικό θα πρέπει να περιλαμβάνονται με αναφορά ε, στις, ε, στους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού ε, Εργασίας όπως 189 για τις ηλικιακές βοηθούς. Αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα λάβει χώρο λοιπόν μια πολιτική συζήτηση στο μέλλον, αλλά εγώ ήθελα να πω ότι δεν θέλουμε την εξαίρεση επουδενή κανενός εργαζόμενου να μην δημιουργήσουμε νομικά κενά και κανείς σίγουρα δεν θέλει να χάσει χρόνο σε, μια, σε ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο ε, θα εξουδετερωθεί στην πράξη, τα μείνει αν περιεχομένου ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η περίοδος ε, εφαρμογής του. Τέλος, θέλω να αναφέρω σε ό,τι αφορά τις προθέσεις μας το εξής. οποιοδήποτε συμβιβασμός ε, επιτευχθεί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη προ, προφανώς της την εθνική νομοθεσία αλλά και τις ε, συλλογικές συμβάσεις, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τους κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι θα πρέπει να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Από τους πρασίνους δεν βλέπω τον κύριο Μέτσερις. Άρα πάμε στην ομάδα EFTT που επίσης απουσιάζει όπως και η ομάδα ENF. Συνεπώς θα πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι που το ζήτησαν. Η πρώτη η κυρία Γιάννη Σλοβέκη. Ευχαριστώ πρόεδρε. όπως και οι προλαλήσαντες, έτσι και εγώ πιστεύω ότι ε, η οδηγία αυτή για τους διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Οι τρόποι εργασία τροποποιούνται, οι όροι εργασία μεταβάλλονται και θα πρέπει να προσαρμοστεί και η κοινοτική νομοθεσία. Ωστόσο, ορισμένες από τις ε, διατάξεις προβλέπονται στην πρόταση αυτής πρόταση αυτή οδηγίας δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το στόχο. Και αναφέρομαι όλος ιδιαιτέρως στους ορισμούς που χρησιμοποιούνται για τις σχέσεις εργασίας, για τον ορισμό που δίδεται για τον εργαζόμενο και τον ορισμό που προβάλλεται για τον εργοδότη. Ξέρετε ότι εδώ η κατάσταση διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Τα κράτη-μέλη έχουν του δικού του άλλωστε ορισμού. Ένα κοινοτικό ενωσιακό ορισμό δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να λειτουργήσει αν δεν λάβει υπόψη του τι υφιστάμενε διαφορέ από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Νομίζω ότι θα προκύψει τελικά ένα νομικό χάο. Και γι' αυτόν τον λόγο, κυρία Μακιντάιερ, και πολύ σωστά είπε ότι θα χρειάζεται εδώ πέρα απόλυτη ακρίβεια. Υπάρχουν τόσο διαφορετικά μοντέλα απασχόληση. Επομένω, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρχουν και πολύ διαφορετικοί ορισμοί όσον αφορά την απασχόληση. Όσον αφορά τώρα του όρου απασχόληση, του όρου εργασία, ξέρετε ότι απαιτείται όλο και περισσότερο ευελιξία. Και αυτό διότι οι εργοδότες αναφέρονται σε κάποιους όρους εργασίας κατά την αρχική συνέντευξη, ενώ η γραπτή σύμβαση που έρχεται στη συνέχεια όχι μόνο φτάνει σε μεταγενέστερο χρονικό στάδιο, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει τελικά και διαφορετικά στοιχεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να προβλέπετε μία ελάχιστη χρονική σε 7 ημερών ανάμεσα στην αρχική συνέντευξη και την ε, γραπτή σύμβαση. Οι γραπτές πληροφορίες για τους αποσπασμένους των εργαζομένους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και θα πρέπει να προβλέπεται τη δυνατότητα να παρακολουθεί κανείς το πόσο διαφανής είναι η ώρα εργασίας σε κυβερνητικά μάλιστα, σε κυβερνητικούς ιστότοπους. όσον αφορά τώρα τους υπόλοιπους τομείς που καλύπτονται από την οδηγία. Αν πραγματικά θέλουμε πιο διαφανείς όρους εργασίας και για την αποσπασμένη εργασία, σαφώς ο στόχος αυτός είναι πολύ θετικός, Απλώς θα πρέπει να αποφύγουμε εδώ πέρα να επαναλάβουμε νομοθετικές διατάξεις που έχουμε σε άλλες οδηγίες, όπως για παράδειγμα στην οδηγία για την ε, προσωρινή απασχόληση. Νομίζω λοιπόν ότι όπου υπάρχουν ήδη ισχύουσες διατάξεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται εδώ πέρα σε αυτή την πρόταση οδηγίας. Προσβλέπω και εγώ σε μια θετική συνεργασία και ελπίζω ότι θα ολοκληρώσουμε το έργο αυτό μέχρι το τέλος της θητείας. Ο κύριος Μπάχτορ έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υπεκρατεί κάποια ομόνια και συνεργασία σε αντίθεση με το εξωτερικό του Κοινοβουλίου, όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ακόμα. Ακούστηκε το θέμα του ορισμού. Παρόλε τι δυσκολίες, νομίζω ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με ειλικρίνεια και παρόλα αυτά να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια λύση έχω επιφυλάξει. Αν δεν το κάνουμε εμεί, κάποια στιγμή θα έρθει να το κάνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και θα πρέπει να έρθει να κάνει τη δουλειά μα και να το νομοθέτει. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο, ούτε σωστό. Οι αυτοαπασχολούμενοι, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να εξαιρούνται από την οδηγία. Βέβαια, να προσέχουμε να μην ε, ενισχυθεί έτσι η στάση των ψευδών απασχολουμένων. Και όπως είπε η κυρία Μάκεντάιρ, να μην επιτρέπονται σχήματα τύπου pay to fly, να πληρώνει δηλαδή ο εργαζόμενος για να εκπαιδευτεί, να κάνει τη δουλειά του. Επίσης, από την πρώτη μέρα θα πρέπει να ξέρει ο εργαζόμενος ποια είναι η διάρκεια της σύμβασή του και το ωράριο του εργασίας. Και όλες οι υπόλοιπε προφορίες το αργότερο μετά από δύο εβδομάδε. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουμε ε, στα πρακτορία ε, που παρέχουν εργασία που είναι κάποιοι μεσάζοντες γιατί δεν έχει επαφή ο εργαζόμενος με τον εργοδότη του. Αλλά όλα αυτά τα ζητήματα της εργοδότησης και των συμβολέων τα διεκπαιρεώνουν κάποιες εταιρείε ενδιάμεσες. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε βεβαίως ε, στην οδηγία το ρόλο των κοινωνικών εταίρων ε, στις εθνικές συλλογικές ε, διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις. Και βέβαια και οι εργασία εργασίας θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν με ρόλο πιο πρωταγωνιστικό και να υπάρχει ε, ασφάλεια δικαίου και επιβολή κυρώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam Ευχαριστούμε κυρία Σόιτροβα. Τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Συμφωνώ ότι όντως θα πρέπει να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, χωρίς όμως να δημιουργούμε νέα εμπόδια και νέου φραγμούς. Έχω καταθέσει ορισμένες σχετικές τροπολογίες και προτείνω να διαγραφεί ο νοσιακός ορισμός προβλέπεται εδώ πέρα. Είμαι υπέρ της δέσμευσης του κυρίου Σαμπόν να καταφέρει να καταλήξει σε μία συμβαστική τέλο πάντων διατύπωση. Ενδεχομένως αυτό να μπορούσαμε να το συστήσουμε περισσότερο. Νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνος ο ορισμός του εργαζόμενου που προτείνεται στην πρόταση οδηγίας. Ενδεχομένως να καταφέρουμε λοιπόν να τροποποιήσουμε αυτό τον προτινόμενο ορισμό. Προφανώς θα προτιμούσα μια καλύτερη εκδοχή του ορισμού αυτού, γιατί θα πρέπει να βελτιωθούν οι όροι εργασία. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τους εργοδότες, για τους εργαζόμενους με συγχωρείτε, αλλά βέβαια και για τους εργοδότες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η βελτίωση αυτή των όρων εργασία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιτευχθεί χωρί τη συμμετοχή των εργοδοτών. Ελπίζω λοιπόν θα καταφέρουμε να κινηθούμε σε αυτό το δρόμο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς για αυτή την πρώτη εισαγωγική συζήτηση. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο ή στους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Όλσον θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε Είναι τιμή και χαρά να δουλεύουμε σε αυτό το θέμα, διότι αυτό δείχνει την ισχύ της ε, διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως θα θυμάστε, μετά την υιοθέτηση του κοινωνικού πυλώνα, η Κομισιόν βιάστηκε να υποβάλει αυτή την πρόταση. Το Συμβούλιο μέσα σε έξι μόνο μήνες κατέληξε σε μια κοινή θέση, σε μια θέση μάλλον, και τώρα βλέπω πως εσείς έχετε προχωρήσει τόσο πολύ. Και με βάση αυτά που ακούω μπορώ να είμαι αισιόδοξο. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Γι' αυτό είμαι περήφανος που δουλεύουμε μαζί. Εκ μέρους του Πρόεδρου Γιούνκερ και της Επιτρόπου Τίσεν που προσωπικά εμπλέκονται, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς, την Επιτροπή, το προσωπικό, για αυτή την ε, προσπάθεια να εμβαθύνετε και να προχωρήσετε γρήγορα. Όπως γνωρίζετε, η κρίση οδήγησε σε μια μεγάλη διαφοροποίηση του εργατικού δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και πολλές εξελίξεις που οφείλονται στην ψηφιακή εποχή. Όλα αυτά οδηγούν σε μια πολύπτυχη και πολυεπίπεδη αγορά εργασίας που είναι δύσκολο να την παρακολουθήσουμε. Οπότε, τι δυνατότητες έχουμε, είτε να δούμε ξεχωριστά μία-μία τις διαφορετικές του διαφορετικού τύπου συμβάσεων ή αυτό που κάναμε εμείς να προσπαθήσουμε οριζόντια να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτής της πολυμορφίας με κοινέ πολιτικές αρχές μέσω ενός κοινού ορισμού, ευρωπαϊκού ορισμού για τον εργαζόμενο κάτι πραγματικά είναι ιστορική σημασίας, είναι ένα παράθυρο, μια ευκαιρία να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο κοινό ορισμό σε, για μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και δεύτερον μια διαφάνεια που θα επιτρέψει ιδιαίτερα στους πιο επισφαλείς εργαζόμενους, ε, τους ε, ποδηλάτες της Deliveroo, ε, τους ε, οδηγούς ε, και που δεν ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, πότε θα πώς θα καταφέρουν να επιζήσουν στους επόμενους μήνες κλπ. Να έχουν ενημέρωση από την πρώτη μέρα που προσλαμβάνονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το θέμα της ενημέρωσης την πρώτη μέρα. Προκειμένου τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα εξ αρχής. Και μετά έχουμε και το θέμα της ε, απαρίθμησης των ελάχιστων δικαιωμάτων για αυτούς τους εργαζόμενου, τους επισφαλείς εργαζόμενου, σε ό,τι αφορά τη δοκιμαστική περίοδο, την επιμόρφωση, την προβλεψιμότητα. Με μετριοπάθεια το κάνουμε βέβαια, προκειμένου να καταπολύσουμε τις πιο σημαντικές ανισορροπίε και καταχρήσει. Ο εισηγητή το αντιμετωπίζει πολύ καλά στο προσχέδιο εκθεσή του και όπω είπε, οι τροπολογίες φαίνεται να οδηγούν προς την κατεύθυνση ενός δίκαιου συμβιβασμού. Δύο θέματα θέλω να σχολιάσω. Ο, το ένα είναι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Στην πρότασή μας προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα ισχυρό ρόλο στους κοινωνικούς εταίρους. Ορισμένα συστήματα κοινωνικών εταίρων βέβαια είναι τόσο ισχυρά ήδη που αυτό που προτείνουμε εμείς ίσως υστερεί λίγο σε σχέση με αυτό που εφαρμόζεται. Πρέπει όμως να βρούμε μια λύση που θα βοηθήσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου ισχυρά κοινωνικά μοντέλα. Ελπίζω ότι ο εισηγητής θα ε, καταφέρει να υποβάλει κάποια πρόταση γι' αυτό. Και δεύτερον, την επικάλυψη με τις ισχύουσες οδηγίες. Είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα με ισχύουσες οδηγίες. Είναι συνεπές το κείμενο αυτό που έχουμε υποβάλει σε ό,τι αφορά το, τα όσα έχουν ήδη προβλεφθεί από άλλες οδηγίες. Παρόλα αυτά, αν χρειάζεται να το εξηγήσουμε περισσότερο, πολύ ευχαρίστως. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι δυνατόν να εμφανιστούν επικαλύψει, αλλά ήδη στο Συμβούλιο Συζήτηση που έγινε δεν εντοπίστηκαν τέτοιου είδου προβλήματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, θέλει κανεί άλλο το λόγο? Ναι, θα επανέλθουμε στον εισηγητή. Παρακαλώ. Θα μιλήσω και στα αγγλικά και στα ισπανικά, ανάλογα στο σε ποιον απαντώ. Θα σχολιάσω πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, γιατί πράγματι ε, από εδώ και πέρα θα εργαζόμαστε επί τη βάση των όσων ε, ελέγχθησαν στις τοποθετήσεις. Στο συνάλφο από το ΕΛΚ, να τον ευχαριστήσω καταρχήν για τα καλά του λόγια και τη στήριξή του. Βέβαια, ασφαλώς είναι σημαντικό όταν νομοθετούμε να είμαστε προσεκτικοί. Η οδηγία αυτή καθορίζει δικαιώματα. Δεν δημιουργεί νομοθετικούς κώδικες. Ούτε σε ευρωπαϊκό ούτε σε εθνικό επίπεδο. Για να πετύχουμε όμως μπορώ να σας ενημερώσω ήδη ότι έχω ξεκινήσει να εργάζομαι με την ομάδα των νομικών, η οποία θα είναι παρούσα στις συνεδριάσεις μας. Και όταν καταλήξουν σε μια συμφωνία μπορούμε να ζητήσουμε τη γνώμη τους για το κατά πόσον είμαστε ασφαλείς από νομικής πλευράς. Σίγουρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την γνωμοδότησή τους. Α, για, το, για τους συναδέλφους από τους σοσιαλιστές. Να σας πω το εξής. Η, στις συναντήσεις μας το ΕΛΚ επέμενε στο εξής. Θα πρέπει οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο κοινωνικός διάλογο οι διαπραγματεύσει που γίνονται στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου θα προστατευθούν και σε ορισμένες χώρες που είναι χώρες μοντέλα η μεταγραφή της οδηγίας αυτής στο νόμο γίνεται μέσω των συλλογικών συμβάσεων και του κοινωνικού διαλόγου α, και αυτό θα πρέπει να τύχει σεβασμού. Θα το υπογραμμίσω ξανά και ξανά και το δέχομαι. Είμαστε ανοιχτοί σε, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε τύπου μεταγραφή στο εθνικό δίκαιο ή ε, στο εθνικό σύστημα τη κάθε χώρα. Αυτό μπορεί να είναι νόμο, μπορεί όμω να είναι συλλογικέ συμβάσει, συλλογικέ διαπραγματεύσει κλπ. Εγώ δεν επιθυμώ απλώς να μην εξαιρεθεί κανένας από αυτούς που έχουν δικαιώματα. Δεν περιορίζομαι στο ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι με ελάχιστες εξαιρέσει ή δυνατόν μηδενική, μηδενικές εξαιρέσεις. Εγώ είμαι ακόμα πιο ριζοσπαστικό. Θέλω να αποφύγω το νομικό dumping. Να το πω έτσι. Τι εννοώ. Δεν θέλω να δώσουμε στις, στα κράτη-μέλη το δικαίωμα μέσω ορισμών να ε, προσδιορίσουν ποιοι καλύπτονται και με αυτόν τον τρόπο να αφήσουν εκτός κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να μείνουν εκτός. Δηλαδή δεν θέλω μια χώρα να μου πει ο οδηγός της Deliveroo δεν είναι εργαζόμενος για μας. Δεν με νοιάζει πώς το ονομάζετε εσείς στον νόμο σας, στην νομοθεσία σας, στις συλλογικές σας συμβάσεις, αλλά αν ο οδηγός της Deliveroo εξαρτάται, βρίσκεται σε μια σχέση εξάρτησης, οικονομικής εξάρτησης, οργανωτικής εξάρτησης, ιεραρχική εξάρτησης κλπ, πρέπει να καλύπτεται. Και πέστε τον εσείς όπως θέλετε μετά, στην εθνική Συνομοθεσία. δεν θέλω να δημιουργήσουμε παραθυράκια μέσω ορισμών σε εθνικό επίπεδο. Καδώστε τους ορισμούς που θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά τα χαρακτηριστικά είναι πολύ συγκεκριμένα και λίγα. Αν είναι ένα φυσικό πρόσωπο που εξαρτάται, σε σχέση που βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης, καλύπτεται. Αυτό θέλω να πω. Να το διακηρύξω προς όλους. Ε, άκουσα με πολύ προσοχή την άποψη της ΓΚΟΕ περί ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της αντιρρήσει ό,τι αφορά το εργαζόμενο να πληρώνουν την επιμόρφωσή τους ε, την κατάρτισή τους. Έχουμε πολλά θέματα στα οποία θα εργαστούμε, δεν θέλω να επισέλθω, επισέλθω σε λεπτομέρειες. Άκουσα και τους συναδέλφους από το ΕΛΚ όχι τον, δεν μιλώ για τον εισηγητή, συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε. Για παράδειγμα την ανησυχία του κ. Μπαχ. Για τους προσωρινούς ε, εργαζόμενους οι οποίοι προσλαμβάνονται μέσω ε, εταιριών αναζήτησης προσωπικού. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας πραγματικά για τις ε, προτάσεις σας και για τις ιδέες σας. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ευαίσθητο το πρόβλημα. Ε, άκουσα την Ντανούτα, άκουσα και τους άλλους συναδέλφους. Χωρίς εργοδότες ασφαλώς και δεν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις. Οπότε είναι σημαντικοί εργοδότες, αλλά όχι μόνο για μένα. Και ήθελα να είμαι ειλικρινής. Είπα, δεν θέλω να έχουμε παραθυράκια, αλλά πρέπει να τους έχουμε υπόψη μας και να μην είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Είναι σημαντική όχι μόνο επειδή υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και σε μεγάλα νούμερα, αλλά θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να κάνουν και καλά τη δουλειά τους, χωρίς βέβαια να καταχρώνται και με σεβασμό στους κανόνες της κοινωνίας. Ευχαριστώ επίσης την Κομισιόν. Είναι τιμή και χαρά είπε η, Κομισιόν να συνεργάζεται μαζί μας και για μας το ίδιο για αυτό το θέμα, αλλά εκτός αυτού είναι και καθήκον μας. καθήκον προς την κοινωνία, προς τους ψηφοφόρους μας, και θα κάνω ό,τι μπορώ, χωρίς βέβαια να υπερβώ τις πεπιθήσεις μου, να βρω ένα συμβασμό. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι πραγματικά σημαντικό, πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αν επιμείνει η Κομισιόν σε ένα ευρωπαϊκό ορισμό των εργαζομένων. Ας αφήσουμε τα δικαστήρια κάθε φορά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να δώσουν έμεσα ένα τέτοιο ορισμό. Διότι αλλιώς αν προσπαθήσουμε τώρα κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας να υιοθετήσουμε ένα τέτοιο ορισμό θα πυροβολήσουμε τον εαυτό μας το πόδια. Ας κάνουμε το πρώτο βήμα και μετά ας αφήσουμε τα δικαστήρια να δώσουν μορφή. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε σε αυτό το σημαντικό μας καθήκον αν επιμείνουμε στον ορισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καλβέ Σαμπον και τους άλλους ομιλητές μας για τη συζήτηση αυτή. Το θέμα είναι πάρα πολύ περίπλοκο αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε και χρονοδιάγραμμα. 18 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Έχουμε ακόμα χρόνο να δούμε τα θέματα αυτά και να ε, βρούμε τους καλύτερους ορισμούς και τις καλύτερες λύσεις. Λοιπόν, τώρα έχει έρθει η ώρα του μεσημεριανού διαλύματος. Μην ξεχνάτε ότι θα τα ξαναπούμε στις 3 το απόγευμα, όχι στις 2.30 όπως είχε αρχικά οριστεί, για να συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus και κάνουμε και το εργαστήρι μας για το θέμα αυτό. Ελπίζω να το θεωρείτε αρκετά σημαντικό και ενδιαφέρον για να έρθετε. Είναι πολλά τα λεφτά και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας αυτό το Ταμείο. Μέχρι τώρα το έχουμε χειριστεί πολύ καλά. Ραντεβού στις 3 λοιπόν. Θα χαρώ να σας ξαναδώ. Για την ώρα χαίρετε και σας ευχαριστώ.